Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καθίστε παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Αρχίζουμε και πάλι τη συνεδρία της Επιτροπής ε, Ντουά που ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί και στην απογευματινή ημερήσια διάταξη έχουμε καταρχήν μία ακρόαση για τον Διαμερικανικό Μηχανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και στη συνέχεια έχουμε μια ακρόαση, όχι ακριβώς ακρόαση, μια ανταλλαγή απόψεων για την Αλγερία. Για την ακρόαση για το Διαμερικανικό Μηχανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας ε, ε, στο βήμα ε, άτομα όλων των ηλικιών και των δύο φίλων και με μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να διδαχθούμε πολλά και να πληροφορηθούμε για, τα, για τις εμπειρίες και το έργο του διαμερικανικού μηχανισμού. Είμαι λίγο απογοητευμένη διότι ο κύριος Γκαρθίας Γιάν, πρόεδρος του Διαμερικανικού Μηχανισμού, είχε καταρχήν δεχθεί την πρόσκλησή μας να έρθει, αλλά μετά μας είπε ότι δεν είχε χρόνο. Τέλο πάντων, μου φάνηκε ότι δεν ήταν πολύ πιστικός ο λόγος που μας έδωσε, γι' αυτό απογοητεύτηκα. Εμεί στην, Επιτροπή, στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν υποστηρίζουμε την α ή τη β πολιτική άποψη. των λεχθέντων θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι ως περιφερειακός οργανισμός και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να εντείνουμε τις σχέσεις μας όχι μόνο σε διμερές επίπεδο αλλά και με περιφερειακές οντότητες και γι' αυτό χαίρομαι που έχουμε εδώ μια ανταλλαγή απόψεων με ένα περιφερειακό οργανισμό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει και η Επιτροπή ΛΥΜΠ ε, που ασχολείται με, τα, με τις ανθρώπινες ελευθερίες και Έχουμε επίσης και ε, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μετά την ε, Λισαβόνα. Από το φθινόπωρο αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα με κάποια κράτη-μέλη που επιβραδύνουν τη διαδικασία της ε, προσχώρησης της Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σίγουρα θα έχετε και εσείς τα δικά σας προβλήματα στη δική σας περιφέρεια. Στην ετήσια έκθεσή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο ζητήσαμε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Επιτροπή να αναλάβουν δράση και θα σας πω τι τους ζητήσαμε στην έκθεσή μας. Τους ζητήσαμε να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες όλων των δικαστηρίων που ασχολούνται με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξετάσουν το ότι πρέπει να δοθεί μέγιστη υποστήριξη στο έργο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών και ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα βήματα για να διευκολυνθεί η δημιουργία ενό ε, δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι χώρε Ασία και Ειρηνικού. Σας έκανα αυτή την παράθεση για να σας δείξω πόσο υποστηρίζουμε τη δουλειά σας, ε, τη δουλειά του Δικαστηρίου και τη δουλειά του της Διαμερικανικής Επιτροπής. Θέλουμε να ε, υπερνικήσουμε την ατιμορρησία. Αυτό είναι ένα μόνιμο ζήτημα προτεραιότητα για μα. Και σε προηγούμενες συναντήσεις καλέσαμε προσκεκλημένους από το Διαμερικανικό Μηχανισμό και πρόσφατα Συζητήσαμε ε, τα αποτρόπια εγκλήματα δολοφονίας ε, φεμινιστριών στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα και μαζί με την Επιτροπή Γυναικών οργανώσαμε μία ακρόαση και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους ε, του Διαμερικανικού Δικαστηρίου και της Διαμερικανικής Επιτροπής που μας εξήγησαν την πολιτική τους για το θέμα. Επίσης γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υποστηρίζει οικονομικά το έργο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου και της Διαμερικανικής Επιτροπής και ελπίζω ότι θα ακούσουμε περισσότερα από τον κύριο Κέρτ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω ο κύριος Σαντιάγκο Καντών είναι εκτελεστικός γραμματέας της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα μας μιλήσει για τις τρέχουσες προκλήσεις της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Καντών, σας καλωσορίζουμε. Στη συνέχεια, ε, ο κύριος Οσβάλντο Τσιριμπόγκα, από το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που τώρα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης που θα μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυρία Μάρτα Ιμπέρο Ντόλα από την ε, πρωτοβουλία της Κοπενχάγης. Ε, το γράφει στο κείμενο στα ισπανικά, όχι μόνο πρέπει να μιλάω αγγλικά, αλλά πρέπει να διαβάζω και ισπανικά. Η κυρία Μάλτα Ιμπέρο Ντόλε, λοιπόν, από την de Κοπενχάγκα για, το, για την ε, Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, η κυρία Χιμένα Ρέιες από την Διεθνή Ομοσπονδία των Ενώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στις παρουσιάσεις τους θα μας μιλήσουν για την προοπτική των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Ενρίκε Σάντσες Φάλκον είναι δικηγόρος του κυρίου Λεοπόλτο Λόπες από την Βενεζουέλα, του οποίου η υπόθεση δικάστηκε από το δικαστήριο το Σεπτέμβριο του 2011. Θα μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση Λόπες Μεντόσα κατά Βενεζουέλας. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά σημεία της συζήτησής μας και καλωσορίζουμε και τον κύριο Γκέρτς από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, επικεφαλής της Μονάδας για τα Μέσα Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλωσορίζουμε και μέλη του Διπλωματικού Σώματος. Έχουμε εκπροσώπους από την Πρεσβεία της Κολομβίας, της Βενεζουέλας, από την Πρεσβεία του Μεξικού και δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος, και από το Περού. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους και από την Βολιβία. Συγγνώμη που τους ξέχασα όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι ότι θα ακούσουμε καταρχήν τους εμπειρογνώμονες που είναι, στο, που είναι προσκεκλημένοι. Θα, στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Επιτροπής ε, και οι βουλευτές και αν θέλουν και τα μέλη της, ε, των διπλωματικών, ε, της διπλωματικής υπηρεσίας να λάβουν το λόγο, μπορούν να λάβουν το λόγο, αλλά ε, έχουμε ένα μέγιστο χρονικό όριο των τριών λεπτών. Εκτός από τα μέλη της, Επιτροπής, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουμε τον κύριο Κόρτες Λάσερ από την Αντιπροσωπεία για το Μεξικό. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Καντών και σας παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την πρόσκληση, τη θερμή πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούν να ε, βγουν από όλη αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δέκα χρόνια πριν ήταν διανόητη αυτή η συνεργασία και δεν υπήρχε δέσμευση μεταξύ των διαφόρων διεθνών οργανισμών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την τελευταία δεκαετία προωθήθηκαν πάρα πολύ τα πράγματα και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Επειδή έχω να κάνω με Ευρωπαίους, θα πρέπει να συγκρίνω το δικό μας σύστημα με το δικό σας. Και τα δύο συστήματα ανέκυψαν με διαφορά πέντε ε, χρόνια. Εμείς ξεκινήσαμε το 59, εσείς λίγο νωρίτερα. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι ότι το, στο αμερικανικό σύστημα υπάρχει μία επιτροπή και ένα δικαστήριο για ε, δύο λόγους. Ε, γιατί όταν μιλήσαμε για το διαμερικανικό σύστημα, κρίναμε ότι υπήρχε η ανάγκη να μην δημιουργηθεί μόνο ένα δικαστήριο. Δηλαδή ακούστηκαν πολλές επικρίσεις και ακόμα ακούγονται σε σχέση με αυτό τον διαχωρισμό. Και γι' αυτό το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξελίχθηκε διαφορετικά. Επίσης, το Αμερικανικό σύστημα έχει πολλές εντολές και λειτουργίες που ε, πάνε πέραν από τις μεμονωμένες αγωγές ή προσφυγές. Υπάρχουν και πολλές άλλες δραστηριότητες και ιδιαίτερα της Επιτροπής το Διαμερικανικό Δικαστήριο καθώς και η Επιτροπή προσπαθεί να επιβάλλει την ένομη τάξη εδώ και πολλά χρόνια. Και τα αποτελέσματα από το 79 και μετά είναι πολύ σημαντικά. Η Διαμερικανική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη καταρχήν τις ατομικές προσφυγές. Λαμβάνουμε 1.500 προσφυγές ετησίως και βλέπουμε ότι αυξάνονται ένα και περισσότερο κατά 10% ετησίως. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την εξέτασή του, στη συνέχεια προβαίνει σε συστάσεις. Εάν όμως το εν λόγω κράτος δεν συμμορφωθεί, τότε η προσφυγή ε, προβάλλεται ενώπιον του αμερικανικού, διαμερικανικού δικαστηρίου. Λάβαμε 18.000 ε, καταγγελίες και από αυτές μόνο 20 έφτασαν στο ανώτατο δικαστήριο, στο δικαστήριό μας, δηλαδή το 1%. Στα πλαίσια αυτών των καταγγελιών προσφυγών υπάρχουν και φιλικοί διακανονισμοί. Γίνονται πολύ φιλικοί ε, διακανονισμοί πριν δηλαδή φτάσουμε σε επίπεδο ε, δικαστηρίου. Ως προς τα ε, ασφαλιστικά μέτρα ή μέτρα προστασίας για να προστατευτούν τα δικαιώματα του ατόμου, εκεί λαμβάνουμε υπόψη πολλές φορές συγκεκριμένες καταγγελίες διότι μπορεί ένας ιδιώτης ε, να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του από παραστρατιωτικές οργανώσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες και κρίνει κατά πόσο θα πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της ζωής του εν λόγω ιδιώτη, του εν λόγω φυσικού προσώπου. Δηλαδή μιλάμε για 50-70 ε, ασφαλιστικά μέτρα ετησίως που λαμβάνονται ως προς την εποπτεία της κατάστασης της χώρες ε, προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο περιφέρειας. Θα θυμόσαστε από το 59 πώς εξελίχθηκε η κατάσταση ιδιαίτερα στην Αργεντινή με την στρατιωτική δικτατορία, στη συνέχεια στην Χιλή με την δικτατορία, τη στρατιωτική δικτατορία του Πινοτσέτ εμείς είχαμε επισκεφτεί αυτές τις χώρες και ήμασταν η πρώτη οργάνωση η οποία προέβησε καταγγελίες γιατί μέχρι τότε ίσχυε ο νόμος της σιωπής. Και δεν θα ξεχάσουμε και στην Αργεντινή τις μαζικές δολοφονίες και εξαφανίσεις ανθρώπων. Επίσης, την Ονδούρα μετά από το πραξικόπημα επισκεφτήκαμε τη χώρα για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά το πραξικόπημα. Όπως ξέρετε γίνονται πολλές ακροάσεις ετησίως όπου λαμβάνουμε πληροφορίες από την κοινωνία των πολιτών για να δούμε πού γίνεται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές φορές ε, γίνονται ακροάσεις για να αποτιμήσουμε την κατάσταση. Και η κοινωνία των πολιτών ε, ενημερώνει την Επιτροπή για την κατάσταση. Έτσι, η Διαμερικανική Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί. Επίσης λαμβάνουμε πληροφορίες και εκθέσεις για χώρες. Ακόμα και αν δεν επισκεφτούμε ορισμένες ε, χώρες. Υπάρχουν, εκεί αναφέρονται επικρίσεις και μας ενδιαφέρει να δούμε πόσο μπορούμε να ε, επιλύσουμε, να διευκολύνουμε καταστάσεις ως προς την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχουν οκτώ τμήματα για ειδικέ καταστάσεις, γυναίκες, παιδιά, αυτόχθονες, ε, φυσικά πρόσωπα, στερούμενα προσωπικών ελευθεριών και ούτω καθεξής. Επίσης, προωθούμε δραστηριότητες και προβάλλουμε ασφαλιστικά μέτρα αναθέμα εκεί που χρειάζεται. Θα προσπαθήσω να προχωρήσω αρκετά γρήγορα γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Καταρχήν ε, προβαίνουμε στην αναγνώριση ευθυνών, απόδοση μάλλον ευθυνών, διότι πολλές φορές αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωρίσουμε τις ε, ευθύνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δολοφονία δεκάδων ατόμων μετά από τη βομβιστική ενέργεια στη Μικτή Επιτροπή Ισραήλ-Αργεντινής, τη δολοφονία του κυρίου Ρομέρο στο Σαλβαδόρ από παραστρατιωτικές οργανώσεις. Αποδόθηκαν ευθύνες στο κράτος του Σαλβαδόρ. Πρόσφατα ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ αναγνώσε τις ευθύνες του ε, για τη σφαγή στο Μοσότε, στο Σαλβαδόρ. Πρόκειται για κάτι το πρωτόγνωρο και πρόκειται για υποθέσεις που άγονται ε, ενώπιον του διαμερικανικού δικαστηρίου για την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί όπου, υπάρχουν, όπου γίνεται παραβίαση και για να ληφθούν μέτρα αποζημίωσης. Επίσης έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις δικονομικού χαρακτήρα. Αυτό αφορά τη Χιλή και το Μεξικό όπου έχει αναθεωρηθεί το σύνταγμα τους. Στην περίπτωση της Χιλής ως προς την ελευθερία του εκφράζεσθε, έχει αλλάξει το Σύνταγμα έτσι ώστε να μην υπάρχει προγενέστερη λογοκρισία όπως έχει γίνει σε περιπτώσεις του τύπου ή και κινηματογραφικών έργων. Επίσης, ε, διαμέσω των φιλικών διευθετήσεων προσπαθούμε να λύσουμε ε, υποθέσεις που άπτονται δύο ε, κρατών. Η περίπτωση Μαρία Νταπένια στη Βραζιλία ε, επιλήθη και γι' αυτό στη Βραζιλία οι γυναίκες που, την χάνουν, ε, που υπόκεινται οικογενειακή βία την χάνουν μεγαλύτερης προστασίας. Αυτό μπήκε στους νόμους, στην νομοθεσία της Βραζιλίας. Το Σαλβαδόρ άλλαξε την πολιτική του σε σχέση με την ε, χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς που πάσχουν από AIDS. Ο πρόεδρος του, της, ε, της ε, Παραγουάης επισκέφθηκε ένα ψυχιατρίο και άλλαξε την νομοθεσία σε σχέση με τις ψυχιατρικές παθήσεις. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Μιλώ για τις δίκες που διεξάγονται σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και 20-30 χρόνια. Το 1992 ήμασταν η πρώτη που είπαμε ότι οι νόμοι επί, περί αμνηστίας δεν ήταν σωστοί. Με βάση αυτή τη νομοθεσία του 92 άρχισαν δύο δίκες που εκδικάστηκαν και από το διαμερικανικό δικαστήριο. Και φτάσαμε σε ε, δίκες σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να ε, λάβει μία απόφαση και το ανώτατο δικαστήριο, Άριος Πάγος του, της Αργεντινής. Και γι' αυτό ακριβώς είχαμε ε, υποθέσεις οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο την Αργεντινή αλλά και το Περού. Οι υποθέσεις που άπτονταν ε, δύο χωρών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σκοτώθηκαν χιλιάδες Λατινοαμερικανοί, εξαφανίστηκαν, πολλοί είναι αγνοούμενοι, πολλοί δεν μπορούσαν να φύγουν από τη χώρα και εξαιτίας τώρα αυτών των υποθέσεων δικάζονται πολλοί και πολλές χώρες της περιφέρειας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ασφάλεια δικαίου. Ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά θα ήθελα να επεκταθώ αργότερα και να μου υποβάλλετε ερωτήσεις, αν το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και συγχαρητήρια για την επιτυχία που είχατε. Ίσως αργότερα στη συζήτηση μπορείτε να μας πείτε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και ίσως εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να σας στηρίξουμε. Τώρα ο κύριος ε, Οσβάλντο Ρουίς Ριμπόγκα. Και εσείς γύρω στα 10 λεπτά έχετε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτή την ακρόαση και βεβαίως θα ε, αναφερθώ σε... θα μιλήσω προσωπικά γιατί δεν εκπροσωπώ το δικαστήριο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι καταρχήν θα μιλήσω για τα προβλήματα που υπάρχουν για την εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου και να κάνω και ορισμένες υποδείξεις για το πώς θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί μας η Ευρώπη έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του δικαστηρίου. Μιλώντας λοιπόν για τις δυσκολίες, για τη συμμόρφωση ως προς τις αποφάσεις του δικαστηρίου, θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου, το 80% των ενταλμάτων αποζημίωσης δεν παρουσιάζουν πρόβλημα. Δηλαδή εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Όταν μιλάμε για περιπτώσεις δημόσιας συγνώμης, ε, υπάρχει συμμόρφωση σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Όμως, σε θέματα όπως ε, η διερεύνηση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι κυρώσεις προς τους υπευθύνους ή η έβρεση των ε, αγνοουμένων, σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι η συμμόρφωση είναι αρκετά χαμηλή. Ε, επίσης, ως προς τις αποζημιώσεις, οι αποζημιώσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία δικαστική πράξη, γιατί πολλές φορές πρέπει να συνεργαστούν πολλά κράτη. Πρέπει να γίνουν νομοθετικές αλλαγές, να ενισχυθούν τα εθνικά θεσμικά όργανα και ούτω καθεξής. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αυτό το χαμηλό βαθμό συμμόρφωσης. Και αυτό έχει να κάνει με την ίδια την οργάνωσή μας, διότι στα πλαίσια της εφαρμογής και της συμμόρφωσης βλέπουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική πίεση από τα ίδια τα αμερικανικά αυτά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να προωθηθεί ένας διάλογος μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής έτσι ώστε να συμμετέχουν και τα πολιτικά όργανα του δικαστήριου μας. Και βεβαίως τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να συμμορφωθούν πρωταρχικά. Θα ήθελα να σας ε, μιλήσω για τους παράγοντες που εδώ υπερισχύουν. Ορισμένες χώρες αρνούνται το δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του δικαστηρίου και θεωρούν ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να αναθεωρήσει την εσωτερική τους ένομη τάξη. Θεωρούν επίσης ότι ένα εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να εγκρίνει, να επικυρώσει αυτές τις αποφάσεις, όπως στην περίπτωση της Βενεζουέλας η οποία μέσω του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου έκρινε μη εκτελεστές τις αποφάσεις μας. Όμως το Μεξικό, το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, αναγνώρισε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα εφαρμογής των αποφάσεών μας. Ένας άλλος ε, παράγων είναι η λανθασμένη χρήση και διάκριση των εξουσιών. Πολλοί θεωρούν ότι η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να επηρεάσει τη νομοθετική. Δηλαδή θεωρούν ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αμερόληπτη. Αυτό που απαιτεί όμως το δικαστήριο είναι ο καθένας να έχει τις εξουσίες του, βεβαίως, άλλο το εκτελεστικό, άλλο το νομοθετικό. Ο καθένας όμως θα πρέπει να ανταποκριθεί με το δικό του χώρο. Δηλαδή, θα πρέπει να εντάξει τις δικαστικές αποφάσεις στην εσωτερική ένομη τάξη κάθε κράτος. Επίσης, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν πολλές φορές να εφαρμόσουν τις αποφάσεις. Δηλαδή, στην περίπτωση του Περού υπάρχει ένα διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο και πολλά κράτη δεν έχουν μια τέτοια δομή νομοθετική και διοικητική που να επιτρέπει τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις. Γι' αυτό οι εθνικές αρχές θα πρέπει να δουν πώς και κατά πόσο μπορούν να συμμορφωθούν. Αυτό αφορά και τα ομόσπονδα κράτη, γιατί πολλές φορές υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων. Ένας άλλος παράγων είναι η, η ίδια η δικαστική πορεία η οποία προσκρούει σε ε, γραφειοκρατικά προσκόμματα και γι' αυτό δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχουν Δηλαδή υπάρχει ένα εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει στις αρχές της δικαιοσύνης να έχουν πρόσβαση σε ε, φάκελους της αστυνομίας ή των ανακριτικών αρχών. Γι' αυτό δεν μπορούν να, γίνουν, να διενεργηθούν σωστά οι έρευνες. Ένας πέμπτος παράγων είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχει σωστός διαχωρισμός και επιμερισμός ευθυνών ως προς την εσωτερική ένομη τάξη. Δηλαδή, στη Χιλή ε, προευλήθη μία εξαίρεση ή αναστολή του νόμου περί αμνηστίας. Όμως η Χιλή δεν προέβαλε τους σωστούς νόμους για να μπορέσει να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτή είναι η σκιαγράφηση των παραγόντων που σας έδωσα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με τρεις μεγάλες ομάδες. Καταρχήν δεν υπάρχει επαρκή γνώση του ενδοαμερικανικού συστήματος, πολιτικές δυσκολίες και οικονομικές δυσχέρειες. Και εδώ περνώ στο δεύτερο τμήμα της εισήγησής μου για το πώς θα μπορούσε η Ευρώπη να συνεργαστεί σε αυτούς τους τρεις μεγάλους τομείς. Για παράδειγμα, ως προς την έλλειψη γνώσης του ενδοαμερικανικού συστήματος θα μπορούσαν να προβληθούν εκστρατείες πληροφόρησης έτσι ώστε και το ίδιο το δικαστήριο να διοργανώσει σεμινάρια. Ε, χρηματοδότηση των ΜΚΟ έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης, ε, ο κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε υπαλλήλους, σε ανώτερους υπαλλήλους, συμμετοχή των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, επίσης προωθώντας δημοσιεύσεις. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να έχουν ως στόχο την γνωστοποίηση του έργου του δικαστηρίου. Μιλώ για τη δημόσια αρχή, για τους δικαστικούς, για τις αστυνομικές αρχές και ούτω καθεξής. Γιατί αν δεν είναι γνωστή μία απόφαση του δικαστηρίου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας. Ως προς τις οικονομικές δυσχέρειες, αυτό έχει αναφερθεί πολλές φορές, διότι το διαμερικανικό σύστημα δεν έχει επαρκείς πόρους για να μπορέσει να φέρει εις πέρα στο έργο του. Γι' αυτό η Ευρώπη μπορεί να συνεισφέρει. Δηλαδή, να κάνετε κι εσείς μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων ως προς τη γνωστοποίηση αυτού του έργου το δικαστήριο πρόσφατα δημιούργησε ένα ταμείο υπέρ των θυμάτων. Αυτό το ταμείο επιτρέπει αρρωγή προς τα θύματα που δεν έχουν ε, επαρκή πόρους για να ε, φέρουν ενώπιον της ε, δικαιοσύνης την υπόθεσή, την υπόθεσή τους. Αυτό αφορά υποθέσεις που αντιμετωπίσαμε στην Κουέστα Ρίκα το Ταμείο αυτό δεν έχει επαρκή σπόρους ακόμα. Επίσης ε, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επισκέψεις ή ακροάσεις σε χώρες της περιφέρειας έτσι ώστε οι ίδιοι οι δικαστές in situ να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες ε, αρχές. Υπάρχουν και πολιτικές δυσκολίες. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να άρουμε αυτές τις δυσκολίες. Θα πρέπει να προωθούμε ακροάσεις σαν αυτήν, σαν την παρούσα, για να ε, μπορέσουμε να μελετήσουμε το διαμερικανικό σύστημα και να δούμε τι γίνεται με διάφορα επιμέρους ε, δικαστικά συστήματα όπως αυτό του Μεξικού. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μία ε, διαφοροποίηση του διαλόγου. Δηλαδή, πολλές φορές χρειάζονται συζητήσεις σε επίπεδο πρεσβειών, ενώ άλλες θα πρέπει να εμπλακούν τα εθνικά δικαστήρια. Δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία θέλει να προωθήσει αυτή την, θέλει να εφαρμόσει μια απόφαση του δικαστηρίου, αλλά πολλές φορές υπάρχουν προσκόμματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε κράτος ε, εκπροσωπείται από την πρεσβεία του. Ίσως εκεί θα πρέπει να προωθούνται και να ασκούνται πιέσεις υπέρ της εφαρμογής ε, μιας απόφασης, δικαστικής απόφασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τις συγκεκριμένες προτάσεις προς το Κοινοβουλίο και την Ένωση. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Μάρτα Ιμπέρο Ντόλα και η κυρία Ρέγες. Νομίζω μαζί θα μιλήσετε. Ε, Σας ε, καλημερίζω και εγώ. Ονομάζομαι Μάρτα Ιμπέρο ε, εργάζομαι στην ε, πρωτοβουλία της Κοπενχάγης για την ε, Λατινική και Κεντρική Αμερική. Πρόκειται για μία πλατφόρμα ΜΚΟ και ασχολούμαστε με την Κεντρική Αμερική περισσότερο και το Μεξικό. Εδώ και 20 χρόνια εργασιών αυτής της ε, πλατφόρμας βλέπουμε ότι στην Κεντρική Αμερική και στο Μεξικό υπάρχουν πολλές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει ατιμορρησία, ανίσχυρο θεσμικό σύστημα αντιμετώπισης της βίας και ένα σύστημα γενικού αποκλεισμού. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δίνει μια τελευταία ευκαιρία στα θύματα για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Και είναι και το μοναδικό σύστημα στο οποίο μπορούν να προσφύγουν τα θύματα. Επειδή στόχος είναι η συνεργασία, πολιτικός διάλογος και εξωτερική πολιτική, δηλαδή να εποπτεύουμε για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής και του Δικαστηρίου. Εάν τα κράτη-μέλη αυτόβουλα και καλόπιστα εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις, τότε δεν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύεται το κράτος δικαίου και μιλάμε για οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ε, ο κύριος Καντών και Τσιριβογκάν μίλησαν για τα δύο αυτά θεσμικά όργανα και εμείς θα θέλαμε να σας δώσουμε, να αναφερθούμε μάλλον ορισμένα παραδείγματα για να σας δείξουμε πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι το σύστημα έμπρακτα στην επίλυση διαφόρων το διαμερικανικό δικαστήριο έχει αποφανθεί σε πολλές υποθέσεις όπως στην υπόθεση που αναφέρθηκε η πρόεδρος ενός φυσικού προσώπου κατά του κράτους του Μεξικού. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει ένα ποιοτικό άλμα σε αυτή την απόφαση ε, λήφθη η απόφαση ενός ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, τα θύματα, οι γυναίκες της Λατινικής Αμερικής ε, χρησιμοποίησαν αυτό το ψήφισμα ε, για να το θεωρήσουν σαν ένα είδος δεδικασμένου. Επίσης, η ύπατη εκπρόσωπος, η Λέδη δηλαδή, ε, Άστον, ε, αποτάνθηκε στο δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτής ε, και στην συγκεκριμένη, στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Ο κύριος Καντών μίλησε και για θεματικές ακροάσεις, για μεμονωμένες προσφυγές στις Ονδούρες, στο Μπαχαγουάν, το Σεπτέμβριο του, από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 σκοτώθηκαν 42 αγρότες μέσα στα πλαίσια του αγροτικού ζητήματος. Μετά από την ακρόασή μας, η Επιτροπή γνωστοποίησε την ανησυχία της για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή την περιφέρεια τότε σταμάτησαν οι δολοφονίες αγροτών σε αυτή την περιφέρεια, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τα δύο τελευταία χρόνια. Ε, δυστυχώς, ο Δον Ματίας Μάρντε, ε, δολοφονήθηκε στο Μπαχαγκουάν. Εν πάση περιπτώσει όμως μειώθηκε η βία Επίσης, συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις. Το ανέφερε ο κύριος Καντών, ιδιαίτερα στο κράτος της Ονδούρας και προβάλλονται και ασφαλιστικά μέτρα καθώς και καταγγελίες για την ε, στρατιωτικοποίηση του Μπαχαγκουάν. Από το Μάιο του 2010 επιτράπηκε σε 18 κοινότητες, Μάιας να μπορέσουν να ακολουθήσουν να αποτελέσουν αντικείμενο ασφαλιστικών μέτρων και αυτό μέσα στα πλαίσια και της λειτουργίας των ορυχείων. Πολλές αποφάσεις άλλαξαν όμως η Γουατεμάλα θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι κοινότητες αυτές να έχουν ε, πρόσβαση στο πόσιμο νερό και να μην υπάρχει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα ορυχεία. Υπάρχουν και άλλα ε, παραδείγματα, σωρία παραδειγμάτων. Όμως το μήνυμά μας είναι ότι το διαμερικανικό σύστημα ε, δημιουργεί ένα ποιοτικό άλμα στην υπεράσπιση θυμάτων και επιβάλλει σε κράτη να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να λάβουν μέτρα. Επίσης, είμαστε υπέρ του, ταχθήκαμε υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του διαμερικανικού συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα μέσω πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας. Η συνεργασία αφορά διάφορα μέσα γεωγραφικού χαρακτήρα, θεματικού. Υπάρχει το ε, Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Μέσο, Μέσο Δημοκρατίας και Ανάπτυξης δηλαδή. Άρα μπορούμε να έχουμε συνεργασία σε περιφερειακό, υποπεριφερειακό επίπεδο, ε, διμερών σχέσεων και βεβαίως και οι αντιπροσωπείες και οι πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προωθήσουν αυτό το διάλογο με τη, ε, τα διάφορα, τις διάφορους κρατικούς φορείς σε επίπεδο αρχηγών κρατών και ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μας ενδιαφέρει να εφαρμόζουν οι αποφάσεις του δικαστηρίου. Στον, ε, ε, στο πλαίσια του Eurolat θα πρέπει να προβλέπονται και επισκέψεις σε τρίτες χώρες. Μπορούμε λοιπόν να προβούμε σε ένα διάλογο και μπορούν μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δει ποιες είναι, ε, ποια είναι η πορεία του συστήματος και οι προκλήσεις για να δούμε ποια είναι και οι απότεροι στόχοι. Μας ενδιαφέρει η υποστήριξη και η χρηματοδότηση, η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και η τεχνική αρρωγή μέσα στα πλαίσια της επίλυσης διαφορών. Να υπάρχει συμμετοχή στις, στην επακροατηρίου ε, διαδικασία, γιατί εάν δεν συμμετέχει η ε, κοινωνία των πολιτών, πολλές φορές η εφαρμογή πέφτει στο κενό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη και σε πρακτικά ζητήματα, δηλαδή βάσεις δεδομένων, χρηστές πρακτικές και ούτω καθεξής. Συμφωνώ με τους κυρίους Καντών και Τσιριμπόγκα για να ε, υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης. Υπάρχει σωρία δυνατοτήτων. Ο κύριος Τσιριμπόγκα μίλησε για διερεύνηση υποθέσεων που οδήγησαν στη βία. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το εσωτερικό δίκαιο, η εκπαίδευση, η αποκατάσταση και ούτω καθεξής. Όπως είπε και ο κύριος Σιριμπόγα, θα πρέπει να υπάρχει και δικαστική αρρωγή των θυμάτων. Εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα θύματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και δεν την χάνουν ε, προστασίας. Γι' αυτό το Ταμείο Υπέρ των Θυμάτων βοηθά στην ε, επίλυση διαφορών. Και θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσουμε τις σχέσεις αυτές και την περαιτέρω διερεύνηση υποθέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τις συστάσεις σας. Τώρα λέει εδώ πέρα, εμένα έλεγε ότι θα μοιραστείτε τα 10 λεπτά. Ε, μακρηγόρησε λίγο συνάδελφος, θα μιλήσω εγώ λίγο λιγότερο. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Μιλήστε, απλά να το ξέρετε. Εντάξει, λεπτά και θα μιλήσω. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, Έχουμε 164 μέλη στον κόσμο και 43 στη Λατινική και Κεντρική Αμερική. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα θέλαμε να μιλήσουμε για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Διαμερικανικού Συστήματος εφαρμογής και μη παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται όμως και πολιτική υποστήριξη. Και αυτό είναι και το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Κατά τους τελευταίους ε, μήνες είχαμε συμφάντα, αρκετά συμφάντα στα πλαίσια κρατών μελών του Διαμερικανικού Δικαστηρίου. Γι' αυτό χρειάζεται υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα της Διαμερικανικής Επιτροπής περί συλλογής γύρω από το θέμα. Πρόκειται για μια ομάδα εργασίας η οποία δημιουργήθηκε για ε, μια πρόσφατη αναθεώρηση η οποία θα πρέπει να προωθηθεί και ο καθένας μπορεί να αποφανθεί. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μην υπάρχουν συστάσεις αποδυνάμωσης. Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες, πολλά κράτη επέκριναν στεναρά το διαμερικανικό σύστημα ε, μιλώντας για λήψη ασφαλιστικών μέτρων που ήταν άδικα και ούτω καθεξής. Πρόκειται για το Περίου, τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία και την Κολομβία. Ιδιαίτερα το, ε, η Βραζιλία και η Κολομβία. Όπως ξέρετε, από το 2001 λήφθησαν ασφαλιστικά μέτρα υπέρ των αυτοχθόνων για να μην δημιουργηθούν οι δικές κατασκευές και εργοστάσια της ε, Μπελομόντε. Θα έπρεπε λοιπόν να ανασταλούν αυτές οι κατασκευές και να αρχίσει μια διαδικασία διαβουλεύσεων με τους ε, αυτόχθονες. Γι' αυτό ζητήθηκε μια μελέτη αντικτύπου. Η Ντίλμα Ρουσέφ, η πρόεδρος, απείλησε να άρει την υποστήριξή της και να ανακαλέσει τον εκπρόσωπο της Βραζιλίας στην Διαμερικανική Επίτροπη. Και δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση, διότι πλήτεται και η αυτονομία της Διαμερικανικής Επιτροπής. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Κατά τη δεκαετία του 90 ε, είχαν ανακύψει και τότε αυτές οι εντάσεις, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη δεν αρέσουν αυτές οι πιέσεις ή οι συστάσεις της Διαμερικανικής Επιτροπής. Στη δεκαετία του 90 μιλούσαμε για δημοκρατική μετάβαση κρατών. Και μιλούσαμε και για φυσικούς πόρους και γύρω από την προστασία των φυσικών πόρων δηλαδή είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη στάση της Βραζιλίας τώρα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να μας υποστηρίξει σε αυτό μας το διάβημα. Δηλαδή να τύχουν υποστήριξης αυτά τα όργανα προστασίας Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν το διαμερικανικό σύστημα. Γιατί θέλουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη στα θύματα παραβίασης. Τον Οκτώβριο του 2011, ο Μανουέλ Σάντος, παρά το γεγονός ότι είχε δεσμευτεί να λάβει μέτρα, έλαβε συγκεκριμένα μέτρα κατά μίας μίκιο και είπε ότι η ΜΚΟ αυτή θα έπρεπε να υποστεί συγκεκριμένες κυρώσεις. Έτσι, Δυστυχώς ε, υπήρξαν πολλές επιπτώσεις. Ε, ξέρετε ότι έγινε μία ε, σφαγή στο Μαπιριπάν όπου το κράτος της Κολομβίας είχε καταδικαστεί το 2006. Ήταν η πρώτη καταδίκη επί παραλήψη, δηλαδή διότι δεν ελήφθησαν μέτρα για να αποφευχθεί αυτή η σφαγή. Δηλαδή οι παραστρατιωτικές, παραστρατιωτικές ε, οργανώσεις εξακολουθούν να δρουν. Δυστυχώς έτσι έρεται κάθε αξιοπιστία μίας μήκυο που είναι πολύ δραστήρια και η οποία εκπροσωπεί τα θύματα τη στιγμή που διεξάγεται μία ε, δίκη και αυτό αφορούσε και εξοδικαστικά μέτρα, όπως είχε πει τότε ο πρόεδρος Ουρίμπε. Επίσης, ε, το δικαστήριο δεν μπορεί να αναγνωρίσει πάντα τα θύματα, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα ε, διερεύνησης in situ. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, τύχουμε της υποστήριξης της κυβέρνησης της Κολομβίας. Σε αυτή την, περίπτωση, την υπόθεση του Ματιριπάν, υπήρχαν έγγραφα στην DAS, στην Υπηρεσία Πληροφοριών, όπου αναφερόταν ότι ίσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπόθεση Μαπυρυπάν για να αποδυναμωθούν οι ΜΚΟ. όπως ε, προαναφέρθηκε, δηλαδή όπως θα μπορούσε να αποδυναμωθεί και η δική σας η ε, υποεπιτροπή. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, λοιπόν και υπάρχει μεγάλη ανάγκη πολιτικής υποστήριξης και ας σταματήσω εδώ. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα συνέρχεται η ομάδα εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων ως προς τις συστάσεις και υπάρχουν πολύ ανησυχητικοί ε, συστάσεις έτσι ώστε να περιοριστεί η ελευθερία του εκφράζεστε. έτσι ώστε να μην προωθούνται και προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην αποδυναμώνονται οι διαφορές. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει με ένα ψήφισμα το Αμερικανικό σύστημα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις δύο περιπτώσεις που μας περιγράψατε. Νομίζω πως αυτό το οποίο θέλατε να είναι να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του δικαστηρίου. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε, γιατί όταν βλέπουμε πως ε, απειλείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από διάφορες χώρες, νομίζω πως είναι παρόμοιος ο μηχανισμός, οπότε είναι κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα της ακρόσης, ε, το τι θα κάνουμε θα το συζητήσουμε. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Φαλκόν, δικηγόρος του κυρίου Λεοπόλντο Λόπεζ από την Βενεζουέλα και θα μας μιλήσει για την περίπτωσή του που εκδικάστηκε στο δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Λεοπόλτο Λόπεφ θα ήθελα να εκφράσει τις ευχαριστίες του διότι ενσωματώσατε την υπόθεση του σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, σε αυτό το διάλογο που ανοίγει μεταξύ α, ε, Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και Ευρώπης. Από πλευράς ε, Λεπόλντο Λόπες ε, και του πολιτικού του φάσματος ανέκυψε μία πολιτική συμμαχία. Χτες προχτές γίναν αυτά. Έτσι ώστε ο κύριος Ενρίκε Ραντόνσκι να μπορέσει να υποβάλει την υποψηφιότητά του και έτσι ώστε ο κύριος Λόπες να μπορέσει να βγει από την πορεία αυτής της ε, σταδιοδρομίας. Εδώ μιλάμε για την υπεράσπιση καθαρά πολιτικών δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα μέσα στα πλαίσια της ευαλωτότητας ε, του δημοκρατικού συστήματος και μέσα στα πλαίσια της ε, καθολικής ψηφοφορίας, η οποία θα έπρεπε να ίσχυε. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που ενυπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα από πλευράς της αντιπολίτευσης των ε, Τσάβες. Το 2008 ο κύριος Λόπες αποτέλεσε ε, θύμα από από πλευράς του ότι δεν μπόρεσε να υποβάλει υποψηφιότητα για τη ε, δημαρχία. Για δημαρχία. Και δεν μπόρεσε φυσικά να εκλεγεί παρά το γεγονός ότι ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της αντιπολίτευσης ήταν υπέρ εκείνου. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να υποβάλει υποψηφιότητα. Υπήρξαν ε, διοικητικά προσκόμματα από μια διοικητική αρχή και αυτό είναι καθαρά αντισυνταγματικό και είναι επίσης τίθεται κατά, μάλλον αντιτάσσεται στην ε, Διαμερικανική Σύμβαση. Δεν μπορούσαν να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση ε, μιλήσαμε, έγινε λόγος και για ε, ποινικά και για ποινικέ κυρώσεις. Επειδή μιλάμε για πολιτικά δικαιώματα, λοιπόν, και ε, δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής, ο κύριος Λόπες προσέφυγε στο διαμερικανικό ε, σύστημα και υπέβαλε αίτημα ενώπιον της Διαμερικανικής Επιτροπής αναλύοντας το θέμα και έφτασε στο συμπέρασμα ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρχε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορούσε δηλαδή να υποβάλει υποψηφιότητα για πολιτικό αξίωμα. Η Διαμερικανική Επίτροπη προσέφυγε με βάση με γνώμονα τις αποφάσεις του δικαστηρίου και προσέφυγε κατά του κράτους της Βενεζουέλας. Όπως ε, καταλαβαίνετε, η απόφαση ήταν ε, θετική, δηλαδή υπέρ του κυρίου Λόπες, διότι ε, παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του κυρίου Λόπες και δεν μπόρεσε να υποβάλει η υποψηφιότητα για πολιτικό αξίωμα. Άρα καταδικάστηκε το κράτος της Βενεζουέλας και ε, κλήθηκε να άρει αυτή την απόφαση. έτσι ώστε να μπορεί το φυσικό αυτό πρόσωπο να υποβάλει η υποψηφιότητα για οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα. Η υποψηφιότητα και η υπόθεση Λεοπόλντο Λόπες είναι ύψης της σημασίας για παρόμοιες υποθέσεις που θα ανακύψουν στο μέλλον, διότι αποτελεί δεδικασμένο Το Διαμερικανικό Δικαστήριο λοιπόν ζήτησε από την κυβέρνηση της ε, Βενεζουέλας να άρει αυτή την απαγόρευση και να λάβει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα έτσι ώστε ο νόμος να μην παραβιάζει αυτό το βασικό δικαίωμα δηλαδή να μην υπάρχουν τέτοια προσκόμματα. Μετά την απόφαση αυτή, είδαμε ε, πολύ μεγάλη λεκτική βία από όλα τα πολιτικά όργανα της Βενεζουέλας, πολιτικά και θεσμικά. Και το συνταγματικό δικαστήριο θεώρησε μη εκτελεστή την απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου λέγοντας ότι είναι ένα αντιδραστικό δικαστήριο και μίλησε για εθνική κυριαρχία. Και γι' αυτό θεώρησε ότι η απόφαση είναι μη εκτελεστή. Άρα δεν υπήρξε συμμόρφωση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου. Ενώπιον όμως της εκλογικής διαδικασίας, δηλαδή οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που προβλέπονται για το 2012-2013, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να χειραγωγήσει την κατάσταση κάνοντας μία προσομοίωση εφαρμογής της απόφασης. Και τι έκανε. Είπε ότι όσοι δεν, υπήρχαν, δεν είχαν εγγραφεί στα εκλογικά μητρώα θα μπορούσαν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Αυτό όμως είναι άκρος αντιφατικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Λόπες δεν, έχει, δεν μπορεί να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Απλώς υπάρχει ένα διοικητικό πρόσκομα το γεγονός ότι είχε προεγγραφεί στα εκλογικά μητρό, στους εκλογικούς καταλόγους και στη συνέχεια λόγω καταδίκης ε, είχε αποσυρθεί το όνομά του. Άρα ε, πρόκειται για ένα καθαρά διοικητικής φύσης ε, πρόσκομα. Τώρα έχει η κατάσταση στην, την παρούσα στιγμή. Δηλαδή, ποια είναι τα διοικητικά προσκόμματα που θέτει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Αυτά είναι πολλά. Και είναι πολλά διότι δεν υπάρχει ε, καταδίκη, δικαστική καταδίκη. Γι' αυτό προβάλλονται διοικητικά προσκόμματα. Γι' αυτό η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να ασκήσει πίεση έτσι ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου να αποφανθεί με βάση ένα ψήφισμα έτσι ώστε στην περίπτωση που ο, ο οποιασδήποτε πολίτης δεν μπορεί να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα, αυτό να μην γίνεται με βάση ε, διοικητικές και διοικητικά προσκόμματα. Πιστεύουμε ότι για να ε, προωθήσουμε ένα δημοκρατικό σύστημα θα πρέπει να αποφανθεί η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να αντιδράσει η Ευρώπη έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Διαμερικανικού Δικαστηρίου. Δεν ξέρω εάν θα ήθελε κανείς ε, περισσότερες εξηγήσεις ε, για το πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστεί μια απόφαση στη Βενεζουέλα σε εθνικό επίπεδο δηλαδή και ακούσαμε και από τη Βραζιλία και άλλες χώρες οπότε θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Γκέτς, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να περιμένετε λίγο για να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές γιατί κάποιοι βιάζονται και θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Εντάξει, ωραία. Και σας διαβεβαιώ θα σας δώσουμε το λόγο αργότερα. Η κυρία Χιμένεθ, λοιπόν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οπωσδήποτε ακροάσεις ε, σαν τη σημερινή είναι πάρα πολύ σημαντικές για να ρίξουν λίγο φως στο διαμερικανικό σύστημα. Υπάρχουν αμφιβολίες στην Ευρώπη για το πώς λειτουργούν αλλού οι μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν σημαντικό να είναι σαφές ε, το εάν οι χώρες ε, στην περιοχή ε, δέχονται τις αποφάσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άκουσα λοιπόν προσεκτικά το πώς η Αργεντινή και η Χιλή ανέτρεψαν τους νόμους περί αμνηστίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Πρέπει τα θύματα να έχουν δικαιοσύνη, πρέπει να λογοδοτήσουν οι εγκληματίες, υπάρχει το δικαίωμα στην αλήθεια, την αξιοπρέπεια. Κάποιος μίλησε για υποθέσεις ε, και το επίπεδο εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις αποφάσεις. Ελπίζω λοιπόν να βελτιωθούν τα επίπεδα συμμόρφωσης Τώρα, τι γίνεται με τις ευθύνες των κρατών μελών όταν μιλάμε για συμμόρφωση με τις αποφάσεις ε, δικαστηρίων. Είναι κρίμα το ότι κάποιες χώρες δεν αποδέχονται τις αποφάσεις. Αυτό το οποίο θα λέγαμε εμείς ως Ευρωπαίοι νομοθέτες είναι να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις χώρες ε, στι χώρε με τι οποίε συναλλασσόμαστε. Εγώ είμαι μέλο αντιπροσωπεία του Μεξικού, όπου ταξιδεύω συχνά, συναντάω τα θύματα, είμαι εισηγήτρια στο Κοινοβούλιο για την οδηγία περί θυμάτων και στήριξη των θυμάτων. Οπότε θα ήθελα να υποστηρίξω τα σχόλια που ακούστηκαν από του ε, ομιλητέ ε, για τη δέσμευση του Μεξικού στην εφαρμογή αποφάσεων ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Γεγονός είναι πως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, θα θέλαμε περισσότερη συνεργασία. Ταξιδέψαμε στην ε, Σιουδά Χουάρες όταν ήμασταν εκεί, συνάντησα πάρα πολλά θύματα που ανισχούν για την ε, προστασία, προστασία τους και γνωρίζω πως η κυβέρνηση του Μεξικού έχει αναγνωρίσει την ευθύνη της σε ορισμένες περιπτώσεις Επίσης εντύπωση μου έκανε το σχόλιο που αφορούσε τη σημασία του διαλόγου, την ανταλλαγή απόψεων. Εγώ είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των θυμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν τακτική ανταλλαγή εκθέσεων, επισκέψεων πρέπει να διατηρήσουμε δεσμούς με αυτές τις χώρες και να μην κάνουμε μόνο ταξίδια στα οποία δεν δίνεται καμία συνέχεια. Πρέπει να είμαστε σε επαφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε μια ε, διοικητική ικανότητα στις ε, χώρες αυτές. Ε, στην διέκθεσή μου το τονίζω αυτό. Όσον αφορά λοιπόν τις χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται με τους διάφορους ε, φορείς ε, του συστήματος. Θα ήθελα να τους ζητήσω να αλλάξουν την ε, πορεία τους. Κυρία Αντεκένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Χωρίς μικρόφωνο κυρία Αντρικένα Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με την ε, κυρία Χιμένεθ όταν λέει πως ε, χαιρόμαστε για το ότι γίνεται σήμερα αυτή η ακρόαση όπως ξέρετε μια αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής μας επισκέφθηκε πέρσι την Ονδούρα και το Μεξικό και πρώτα απ' όλα θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω και εγώ να πω πως χαίρομαι ιδιαίτερα για την ακρόαση αυτή. Ε, να το ακούσει λοιπόν πέρσι μία αποστολή της Επιτροπής μας επισκέφθηκε το Μεξικό και την Ονδούρα. Ο κύριος Κάντσον ανέφερε την Ονδούρα θα ήθελα λοιπόν εσείς να αξιολογήσετε την κατάσταση, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις ε, συναντήσεις μας στη χώρα αυτή, τη συνάντησή μας με τον Υπουργό, την Υπουργό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, η οποία ανέφερε τα προβλήματα του καθεστώτος των δικαστών στη χώρα ε, των δικαστών που δεν υποστήριξαν την αλλαγή της κυβέρνησης το 2009 οι οποίοι απολύθηκαν. Ξέρετε κάτι σχετικά και η Κομισιόν έχει κάποιες ε, σύστασεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίση που έχουμε τον κύριο Σάντσες Φαλκόν εδώ μαζί μας. Στην δε περίπτωση Λεοπόλτο Λόπες δεν ξέραμε εδώ και καιρό, θέλαμε να τον δούμε σήμερα, αλλά βεβαίως για διάφορους λόγους. Η ακρόαση αυτή λαμβάνει χώρα μόλις σήμερα. Χτες η πρεσβεία της Βενεζουέλας έστειλε μια εξήγηση σε μένα και σε άλλους συναδέλφους για το γιατί η απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται και λένε τα ίδια πράγματα που λέτε και εσείς πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σα άποψη γιατί εκπροσωπείτε την Επιτροπή. Πώ αντιδράτε ε, όταν μια χώρα λέει ότι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση. Τι κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση. Και τελευταία παρατήρηση, όχι ερώτηση. Εμείς δεν γνωρίζουμε ολόκληρη την... Κοιτάμε ολόκληρη την περιοχή και βλέπουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Υπάρχει το Μεξικό το οποίο επισκεφτήκαμε και εκεί ακούσαμε σε διάφορες συστάσεις για τις αποφάσεις του δικαστηρίου που εφαρμόζονται με δυσκολίες αλλά εφαρμόζονται σε άλλες περιπτώσεις κάποιες χώρες λένε πως δεν θα εφαρμόσουν αυτές τις ε, αποφάσεις οπότε όπως είπα βλέπουμε πως ε, είναι μια περιοχή με μεγάλες διαφορές ε, από χώρα σε χώρα και αν η υποεπιτροπή μας σύνεται σε ένα έγγραφο νομίζω πως θα ήταν κάτι το λογικό αυτό Σας ευχαριστώ κύριος Μάιερ Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από τα μέσα που έχουμε, δηλαδή τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία, τη Eurolat, να ενισχύσουμε το διαμερικανικό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει και δικαστική αρρωγή των θυμάτων. Αυτό είναι ύψιστη τη σημασίας, αν και είναι δύσκολο. Όπως ξέρετε, ο δικαστής Γκαρθών ε, βρίσκεται στο ε, ε, εδόλιο του κατηγορουμένου γιατί βοήθησε τα θύματα του φραγκισμού. Όπως ξέρετε, στην Αργεντινή δεν υπάρχει παραγραφή, αλλά στην Ισπανία ναι. Στην Ισπανία υπάρχει. Τι να πω, από πλευράς Ευρώπης θα πρέπει να συνεισφέρουμε και εμείς για την ενίσχυση αυτού του διαμερικανικού σύστηματος ε, απόδοσης δικαιοσύνης. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα διότι το ε, διαμερικανικό σύστημα εξαρτάται από το ε, διαμερικανικό δικαστήριο και την Επιτροπή και ίσως με την νέα αυτή δομή συμμετέχουν και είπα. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει. Πιστεύετε ότι κάτι θα αλλάξει έτσι ώστε να υπάρξει μία νέα ε, οργάνωση ή ε, δομή, δηλαδή τη ΣΕΛΑΚ. Έχουν μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη σημασία η μαρτυρία σας και ως προς τα βασανιστήρια, ε, τις εξαφανίσεις και τις δολοφονίες, όλα αυτά μας σοκάρουν όλους και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει ατιμορρησία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο καταπατούνται και πού τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή να δούμε πού αλλού υπάρχουν που αλλού γίνονται ε, δολοφονίες, που γίνονται πραξικοπήματα, που γίνονται βασανισμοί. Δηλαδή, έχετε εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις. Στην ε, περίπτωση της Ονδούρας υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία για την απόδοση ευθυνών στους ε, πραξικοπηματίες. Σε σχέση με τις μαρτυρίες που, στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Φαλκόν. Από, από όσο ξέρω, στη ε, Βενεζουέλα ε, υπάρχει διαδικασία ε, μη αποδοχής για συγκεκριμένους αξιωματούχους και αυτό αφορά ένα 45% για την αντιπολίτευση και 50 κάτι για αξιωματούχους της, της ίδιας της κυβέρνησης. Ο κύριος Λόπες Μεντόσα δεν μπορούσε να συμμετάσχει για συγκεκριμένους λόγους. Πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι υποστήριξε το πραξικόπημα το 2002, γιατί μιλάμε για έναν πραξικοπηματία. Όμως ε, δέχτηκε 60 εκατομμύρια μπολίβαρ, δηλαδή υπεξαίρεσε δημόσιο χρήμα και όταν ήταν δήμαρχος του Τσακάου ε, υπεξαίρεσε χρήματα από τον δημόσιο προϋπολογισμό. Και αυτό δεν είναι λίγο. Πρόκειται για σφετερισμό και υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος. Εχθές βεβαίως αποφάσισε να μην υποβάλει υποψηφιότητα. Ξέρετε πώς έχει η αντιπολίτευση στην Βενεζουέλα. Αυτό είναι δικό του θέμα. Όμως το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας ε, κατέστησε σαφές ότι έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή και του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Άρα γι' αυτό είπε ότι είναι μη εκτελεστή απόφαση διότι έτσι κι αλλιώς του έχουν αποδοθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, άρα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα. Αν δεν θέλει είναι δικό, δική του υπόθεση. Αλλά μπορεί να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα και του εκλέγει και του εκλέγεστε. Μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα αν το επιθυμεί αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα γιατί δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα από όσο γνωρίζουμε. Αυτό το είπα γιατί έχει σημασία. Βεβαίως θα υποστηρίξουμε ως Ευρωπαίοι αυτή τη ε, συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο και μέσα στα πλαίσια της ε, Eurolat έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα χώρο συζήτησης και διαλόγου για να ενισχύσουμε αυτά τα θεσμικά όργανα για την ε, δικαστική εποπτεία ως προς την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Μάγερ και έχω τώρα αρκετούς ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι τις 5 αλλά ας μην ξεχνάμε ότι μας πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος Ομπιέρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το σύνολο των παρεμβάσεων. Είναι όλες πάρα πολύ χρήσιμες ε, για εμάς. Και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μία ορατότητα, αν μπορώ να το πω έτσι, του ε, διαμερικανικού συστήματος για να δούμε ε, κατά πόσο υπάρχει ε, θέμα υλικοτεχνικής υποστήριξης και κατά πόσο μπορούμε να σας υποστηρίξουμε γενικότερα, ενισχύοντας τη συνεργασία. Θα ήθελα όμως εντάχει να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο έφυξε η κυρία Ρέγες για μια υπόθεση στην Κολομβία που με απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, δηλαδή την περίπτωση του Χωσέ Αλβάρε Τρέπο. Πρόκειται για ε, έναν σύλλογο δικηγόρων του δικηγορικού σύλλογου και δεν ξέρω κατά πόσο έχει υποβληθεί σωστά, έχει σκιαγραφηθεί σωστά το θέμα, αλλά θα ήθελα να πω τα εξής. Νομίζω ότι υπάρχει μία στρατηγική αμφισβήτησης προσώπων για να αρθεί η αξιοπιστία του ίδιου του συστήματος, του διαμερικανικού συστήματος ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Και θα ήθελα οι, οι κύριοι Κατών και τσιριβόγκαν να προβούν σε μία αποτίμηση αυτής της κατάστασης. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Όβιολης. Ο κύριος Κόρτες Λάστρο, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Μεξικού. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, διότι οι συνάδελφοι με κάλυψαν εμπολής. Η κυρία Χιμένεθ Μπεθερίλ αναφέρθηκε στην ε, κατάσταση των θυμάτων, αλλά και ο κύριος ε, Ρουίς Τσιριμπόγκα σε σχέση με τον ρόλο μας στις διάφορες αντιπροσωπείες για να μπορέσουμε να εργαστούμε υπέρ ενός διαλόγου. Μέσα στα πλαίσια της Μικτής ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με το Μεξικό συνεργαζόμαστε και στο Μεξικό στην τελευταία συνεδρίαση ανοίξαμε, προωθήσαμε έναν διάλογο και όταν φτάσαμε στα συμπεράσματα, φτάσατε στα συμπεράσματα της έκθεσης, συμμετείχαμε και εμείς. Μετά από τη μετάβασή σας, δηλαδή στο Μεξικό. Προωθήσαμε λοιπόν το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό. Ήταν ένας ανοιχτός διάλογος ένας εκτενής διάλογος και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ζητήσω καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αντιπροσωπιών και επιτροπών για την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες που επισκεπτόμαστε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ακούσαμε τους βουλευτές. Βλέπω πως οι δύο πρέσβεις ζήτησαν το λόγο. Σας ευχαριστώ, αλλά να θυμάστε πως έχετε τρία λεπτά ο καθένας. Πρώτα απ' όλα ο πρέσβης, ο κ. Γκαρσία της Βενεζουέλας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι γιατί θα ήθελα να σας ζητήσω περισσότερο χρόνο για να αναφερθώ στην περίπτωση του κυρίου Λόπες. Γιατί πρόκειται για μία άκρος ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μία από τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά αυτά όργανα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η χρήση που γίνεται για την καταπολέμηση προοδευτικών κυβερνήσεων της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα για την υποψηφιότητα ενός φυσικού προσώπου και για τη χειραγώγηση της ε, πληροφορίας. Δηλαδή λέγονται μισές αλήθειες ή ψεύδι. Και λέγεται ότι ο κύριος ε, Λόπες δεν έχει πολιτικά ε, δικαιώματα. Το 2002 ο κύριος Λόπες συμμετείχε σε ένα κρατικό εθνικό πραξικόπημα και δημιούργησε και φασιστικές ταξιαρχίες και είχε ε, παραβιάσει τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, διότι έβαλε στη φυλακή και πολλούς ε, αντιφρονούντες τότε. Μετά από την ε, πράξη αμνηστίας και την πολιτική σταθεροποίηση της χώρας, που σήμερα γνωρίζουμε, άλλαξε άρδιν η κατάσταση. Είδαμε λοιπόν ότι ο κύριος Λόπες ως εκπρόσωπος ενός πολιτικού κόμματος μπόρεσε να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους για να συμμετέχει στις εκλογές, αλλά χτες απέσυρε την υποψηφιότητά του ως εκπρόσωπος της άκρας δεξιάς στη Βενεζουέλα. Ε, λυπούμεθα διότι υπήρξε ε, μεροληπτική παρουσίαση. Οι νομικοί επίτροποι θεωρούν ότι η απόφαση του διαμερικανικού δικαστηρίου είναι μη εκτελεστή, διότι ο κύριος ε, Λόπες χαίρει των πολιτικών του δικαιωμάτων. και γι' αυτό η απόφαση αυτή δεν μπορούσε να υπερβεί, δηλαδή να υπερισχύσει των εθνικών νόμων. Και γι' αυτό δεν δεχόμαστε αυτή τη θυματοποίηση πολιτικών προσώπων οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διαφθορά και για σφετερισμό του δημοσίου χρήματος, πέρα από το αποτυχημένο πραξικόπνα του 2002. Ευχαριστούμε, κύριε Πρέσβη. Νομίζω πως αναφερθήκαμε σε διάφορες χώρες, λιγότερο ή περισσότερο προοδευτικές, οπότε δεν ήταν απόπειρα να παλέψουν μια προοδευτική κυβέρνηση στη Λατινική Αμερική, γιατί αναφέρθηκαν πολλές φορές και παρόμοια πράγματα έχουμε και στην Ευρώπη. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρεσβευτή της Κολομβίας, τον κύριο Ριβέρα, επίσης για τρία λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητά μέλη της έγκριτης αυτής Επιτροπής, θα Ήθελα να αναφερθώ και εγώ στην υπόθεση Μαπυρίπαν στην ε, Κολομβία και θα ήθελα να σας πω ότι μετά από απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου το 2005 ως αντιστάθμιση και αποζημίωση θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να δούμε τι έγινε με τα θύματα του 97 τα οποία σφαγιάστησαν καθώς και η οικογένειά τους. Με βάση αυτή την απόφαση του Διαμερικανικού ε, Δικαστηρίου, η εισαγγελική αρχή που είναι αναξάρτητη από το εκτελεστικό θεώρησε το Οκτώβριο ότι ο κύριος Ροντρίγες, ε, Μαρτίνες Κορτέιρας και Γκο Φερνάντες, Μαρτίνες Κορτέρας δεν θεωρούνται ε, δίκτυμα με, ε, θύματα με βάση την απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου. Δηλαδή, το Κολομβιανό κράτος και το Διαμερικανικό Δικαστήριο, μάλλον το Διαμερικανικό Δικαστήριο έφτασε σε μία ακρόαση στις 23 του παρελθόντος ε, ε, μηνός και μίλησε για τα θύματα τα οποία ε, δεν μπόρεσαν να εισακωστούν. Μα αυτό το όρισε η εισαγγελική αρχή και όχι η κυβέρνηση της Κολομβίας. Αυτό δημιούργησε μεγάλο σκάνδαλο στην Κολομβία και οι κρατικές αρχές Ε, θεωρήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση αυτού του καθεστώτος και ζητήσαμε από την εισαγγελική Αρχή να διασαφίσει τα θέμα, το θέμα αυτό. Ε, στις 23 του παρελθόντος ε, ζήτησε, ζητήθηκε να διασαφιστεί το ζήτημα έτσι ώστε να το δούμε να ειδωθεί κατά την επόμενη συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Γιατί δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί να θεωρείται κανείς ε, διαφθορέα στη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, εμείς ε, καλή την δράσαμε και ε, η εισαγγελική αρχή έδρασε ξεχωριστά. Εμείς δεν αρνούμεθα τα γεγονότα του 97 στο Μαπυρίπαν και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντισταθμίσουμε αυτή τη βλάβη προς τα πραγματικά θύματα του 97. Θα πρέπει να γίνει αυτή η διευκρίνηση και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πολιτική θέληση να υποστηρίξουμε ως κράτος της Κολομβίας το διαμερικανικό δικαστήριο και την Επιτροπή για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την Ήπειρο. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Και τώρα σύντομα υπάρχει ένα αίτημα παρέμβασης από τον κύριο Μέγκα της ε, Μεξικανικής Πρεσβείας. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, ε, και εμείς ε, έχουμε δράσει σε αυτά τα πλαίσια και χαιρόμαστε για την πρόσκληση για να μπορέσουμε να θίξουμε τόσο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την υποεπιτροπή. Ο πρέσβης δεν μπόρεσε να παραστεί, αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι υποστηρίζουμε το διαμερικανικό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως έχουμε εκφράσει σε πολλά φόρα και είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του συστήματος. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκαν και οι συγητές. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναγνώριση των δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια των εθνικών και διεθνικών οργανώσεων. Προσπαθούμε να δράσουμε μέσα στα πλαίσια της Διαμερικανικής Σύμβασης έτσι ώστε να αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των δικαστικών αρχών. Το Μεξικό τάσεται υπέρ αυτού του μηχανισμού υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευχαριστούμε πολύ και τη Μεξικανική κυβέρνηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε τον κύριο Γκέρτς από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πέντε λεπτά θα σας δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λόχμπιλερ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και είναι κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί σίγουρα το θέμα αξίζει πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω μέσα στα πέντε λεπτά να αναφέρω έξι σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι θέλω να τονίσω την υψηλή σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην εξέταση, λεπτομερή εξέταση που γίνεται για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιφερειακό επίπεδο σε διάφορες χώρες. Και γι' αυτό Υποστηρίζουμε το διαμερικανικό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και επιπλέον αυτής της υποστήριξης έχουμε ε, και μια επιπλέον αγάπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ανέφερε και ο κ. Καντών γιατί το πανευρωπαϊκό σύστημα και το διαμερικανικό σύστημα είναι, ε, έχουν μια αδελφική σχέση ε, γεννήθηκαν και αναπτύσσονται παράλληλα στις δύο υπήρους η αδίποτε μορφή συνεργασίας λοιπόν ε, και γόνιμου διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού και του Αμερικανικού ε, Μηχανισμού είναι ιδιαίτερα θετικό και παράλληλα ε, χαιρετίζουμε και το Αφρικανικό σύστημα και το σύστημα Ασίας και Ειρηνικού που βρίσκεται σε εμβρική μορφή ακόμη η υποστήριξή μας έχει λάβει διάφορες μορφές. Η Μαρία Ριμπέιρο ανέφερε τα βασικά σημεία, πολιτικός διάλογος, διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με χώρες όπως το Μεξικό και η Κολομβία, των οποίων ακούσαμε παρεμβάσεις από τις πρεσβείες. και για την οικονομική συνεργασία και για αυτά που έχει αναφέρει η Λαδιά Άστον. Είναι σημαντική η πρόκληση της επιβολής των αποφάσεων του δικαστηρίου και των προσωρινών μέτρων και άλλων συστάσεων της Επιτροπής. Κατανοούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, κατανοούμε τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, κατανοούμε τον πολύπλοκο χαρακτήρα ε, στην ε, εφαρμογή αυτών των ε, αποφάσεων και συστάσεων. Πολύ σωστά η κυρία Λόχμπιλε αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή εμπειρία, γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες αυτές και υπάρχουν ε, και πολύ γνωστές περιπτώσεις όπως αυτές που ανέφερε η κυρία Ρέγες και σχολίασε και ο πρέσβης της Κολομβίας και άλλες υποθέσεις που είναι γνωστές. Γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά την κατάσταση. Εκεί που ανησυχούμε είναι όταν η διαφορετική ερμηνεία της εφαρμογής οδηγεί σε περιπτώσεις όπου η ακαιρεότητα, η ανεξαρτησία της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου αμφισβητούνται και η ακαιρεότητα και η ανεξαρτησία αυτών ιδίως ε, ε, σε σχέση με τη δυνατότητα συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών με το δικαστήριο. Αυτό μας ανησυχεί, διότι δεν θέλουμε να υπονομευθεί ένα τέτοιο διαμερικανικό σύστημα ή αντίστοιχα δεν θέλουμε να υπονομευθεί και το ευρωπαϊκό σύστημα που έχουμε. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε τέτοιο σημείο, ανησυχούμε. Το επόμενο σημείο μου αφορά την κοινωνία των πολιτών που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, ε, Αμερική, στην υποστήριξη του διαμερικανικού μηχανισμού, λόγω της πρόσβασης ε, στο δικαστήριο και στην Επιτροπή και για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και για την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών πάντοτε στον πολιτικό διάλογο και στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών και οικονομικά υποστηρίζουμε ε, με το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ήταν το τέταρτο σημείο μου και το πέμπτο σημείο αφορά τους οικονομικούς πόρους. Ο συνάδελφος από την ΤΕΦΚΟ είναι εδώ παρόν, ή συνάδελφος μάλλον, και έχουμε συντονισμένες ενέργειες ε, με την ΤΕΦΚΟ Βέβαια έχουν ε, άμεση ευθύνη τα ίδια τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν ε, επαρκώς το Δικαστήριο και την Επιτροπή, γιατί αυτή είναι η κύρια ε, αρμοδιότητά τους. Βέβαια, ήδη από το 2005 και μέχρι σήμερα και μέχρι το 2011-2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα για να προωθεί ε, τέτοιες υποθέσεις που έχουν σχέση με την ελευθερία έκφρασης ε, και για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εξετάσει και εναλλακτικέ μορφές χρηματοδότησης και μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για την Πρόθεση Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έκτο και τελευταίο σημείο αφορά τον πολιτικό διάλογο. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν το 2009 υπέγραψαν ένα, ένα προσύμφωνο ε, και το Φεβρουάριο θα γίνει ο πρώτος πολιτικός διάλογος ε, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σημαντικά ε, αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει και το διαμερικανικό σύστημα μαζί με τον OAS, τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών για να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των άλλων οργανισμών. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ιδιαίτερη σημασία στο να έχουμε ένα μια εξειδικευμένη συνάντηση και διάλογο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Γκέρτς για τις πληροφορίες που μας δώσατε και νομίζω πολλές καλές πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Τώρα κατάλαβα πως δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, τα οποία όμως δεν απευθύνονται σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα, λοιπόν, κύριε Φαλκόν, σύντομα να απαντήσετε στα ερωτήματα του κυρίου Λόπες. Και μετά θα ζητήσω τον κύριο Φαλκόν να επανέλθει στα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα δεν πρέπει να ανοίξουμε γενική συζήτηση. Κύριε Φαλκόν, εσείς πρώτα. Θα ήθελα να πω ότι μιλάμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό αμφισβητείται. Μπορούμε να μιλήσουμε για μία υποκατηγοριοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οριακά. Μιλάμε για καταπολέμηση απολυταρχικών καθεστώτων για να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, να μην ανακύψουν τέτοιες καταστάσεις και στο μέλλον. Έγινε λόγος για διαφθορά. Θα ήθελα να πω όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε μία χορηγία σε μία ΜΚΟ και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι υποψηφιός προς την υποψηφιότητα και τα διοικητικά προσκόμματα δεν έγινε ε, δικαστική έρευνα γιατί δεν υπήρχε λόγος. Μιλάμε για 8-10 χρόνια πριν. Ποτέ δεν παραπέμφθηκε στη ε, δικαιοσύνη ο κύριος Λόπες για κάτι τέτοιο. Τώρα, εάν είχε υποπέσει σε άλλο παράπτωμα κάποια άλλη στιγμή, δεν το ξέρω. Αλλά, εν πάση δεν ε, έγινε δικαστικός αγώνας. Μιλήσατε για 60 εκατομμύρια μπολίβαρες. Όμως δεν αποδείχτηκε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Δεν χρησιμοποίησε δηλαδή αυτό το μηχανισμό ε, στον οποίο αναφορθήκατε εσείς. Δεν έγινε δηλαδή υπεξαίρεση χρήματος. και αναφέρεται ρητά διότι δεν υπήρξε καμία ε, υπόθεση διαφθοράς. Και εδώ μιλώ μόνο για τον κύριο Λόπες. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι ε, που υπάρχουν υποψήφοι που χαίρουν πολιτικών δικαιωμάτων αλλά εδώ πρόκειται για μία ε, σοφιστία καθαρά γιατί μιλάμε για ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο αναφέρει κάτι και για μία απόφαση η οποία αφορά τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας αλλά τη μη δυνατότητα άσκησης των εξουσιών αυτών εάν εκλεγεί κάποιος το αξίωμα αυτό. Ως προς τα στατιστικά στοιχεία η Ναι, βεβαίως ε, πρόκειται για, ε, για υψηλά στατιστικά στοιχεία που αφορούν και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ε, μπορούν να, υπάρχουν, να υπάρχει όμως και χειραγώγηση αριθμητικών στοιχείων όπως θέλουμε. Μπορούμε να μιλάμε για 80% αντιπολίτευση ή 20% συμπολίτευση, αλλά πάντα υπάρχει χειραγώγηση στοιχείων. Δεν υπάρχει δεν υπάρχουν ε, τέτοια στοιχεία τα οποία να μπορούν να ε, ε, αποδειχτούν. Ο κύριος Καντών. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω στις ερωτήσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως μου ζητάτε. Ως προς το θέμα της Ονδούρας υπήρχαν δύο θέματα. Για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, θα ήθελα να πω ότι ξέρουμε ότι στην Ονδούρα έγινε ε, πραξικόπημα τη στιγμή που κάποιος μπαίνει, στρατιωτικοί μπαίνουν στο σπίτι ενός ε, προέδρου, τον βγάζουν από το σπίτι του, τον βάζουν σε ένα αεροπλάνο και το στέλνουν αλλού, ε, έχει γίνει πραξικόπημα, πώς αλλιώς να το πούμε. Υπ' αυτή την έννοια είχαμε ορισμένους δικαστικούς υπαλλήλου οι οποίοι αντιτάχθηκαν σε αυτό και υπέστησαν κυρώσεις για άλλους επιλύθηκε το θέμα και για άλλους όχι. Τα γεγονότα είναι όπως σας τα περιέγραψα πάντως. Και η Επιτροπή μίλησε για ατιμορρησία σε σχέση με τους ε, πραξικοπηματίες που συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Δεν έγιναν σοβαρές έρευνες και δεν τους επιβλήθησαν κυρώσεις. Πολλές φορές μάλιστα ανέλαβαν και σοβαρά πολιτικά και μία αξιώματα. Η αντίδραση της περιφέρειας ήταν θετική. Υπήρξε δηλαδή μια σοβαρή αντίδραση από όλες τις ε, χώρες της περιφέρειας. Ως προς το θέμα της ΣΕΛΑΚ, θα ήθελα να πω ότι σήμερα εάν λάβουμε υπόψη το πολιτικό και το δικαστικό κεκτημένο, οποιαδήποτε αλλαγή γίνει, θα γίνει με βάση τα δεδικασμένα και το κεκτημένο που υπάρχει στα πλαίσια του ε, διαμερικανικού δικαστηρίου. Είναι κάτι που δεν είναι καθόλου απλό βεβαίως. Ως προς την Κολομβία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη ε, ε, διότι μας υποστηρίζει αυτό αφορά και το Μεξικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, ε, πρέσβη του Μεξικού που υποστηρίζεται το διαμερικανικό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε σχέση με το Μαπιριπάν θα ήθελα να πω ότι το διαμερικανικό σύστημα βασίζεται σε πληροφορίες από τα ε, εμπλεκόμενα μέρη. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε έρευνα από μόνοι μας. Στην περίπτωση λοιπόν του Μαπυριπάν, οι πληροφορίες που λάβαμε και στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο για τα θύματα και μετά οι έρευνες που έγιναν βασίστηκαν σε πληροφορίες της Γενικής Εισαγγελίας. Και με βάση αυτές τις πληροφορίες που λάβαμε και από τις Κολομβιανές αρχές, είδαμε ποιοι ήταν θύματα και ποιοι όχι. Και εδώ έδρασε και η εισαγγελική αρχή. Εάν δεν ήταν θύματα, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν θύματα που να αποζημιώνονται που να μην υπήρξαν πραγματικά θύματα. Θα πρέπει λοιπόν να αποσαφινιστεί η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μας έφεραν οι κολομβιανές αρχές και με βάση αυτές δράσαμε. Μιλάμε για ένα, μιλήσατε για ένα σύστημα αναθεώρησης αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση θα πρέπει να διευρύνει την υπεράσπιση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν νέα μέσα και να μην υπάρχουν συσταλτικές ερμηνείες και περιορισμοί. Ως προς την πρώτη παρουσίαση, τη συμμόρφωση και την εφαρμογή, αυτό είναι ένα θέμα ύψης της ε, σημασίας. Μιλάμε για συμμόρφωση, για ποσοστό συμμόρφωσης που είναι αρκετά χαμηλότερο από ό,τι θα θέλαμε, αλλά ως προς ε, ε, τις συμβολικές αποφάσεις βλέπουμε ότι αναθεωρούνται οι νομοθεσίες εκεί που πρέπει. Επίσης υπάρχει χρηματική αποζημίωση και απόδοση ευθυνών, απονομή ευθυνών στα κράτη. Εκεί που δεν υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης πρόκειται για τις προσφυγές των φυσικών προσώπων, τις μεμονωμένες προσφυγές. Εδώ δυστυχώς δεν ε, μπορούμε να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως θα θέλαμε. Υπάρχει μία διαροφοροποίηση και πολλές φορές δεν υπάρχει ε, σωστή και επαρκής επικοινωνία, ιδιαίτερα σε σχέση με την επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Συστήματος με το Διαμερικανικό. Και εδώ μιλώ για το πρόσφατο παρελθόν της ε, περιοχής αυτής. Πλήρη συμμόρφωση θα υπάρχει όταν δεν θα εξαρτώμεθα από την πολιτική θέληση των κυβερνήσεων. Και αυτό θα το κατορθώσουμε όταν υπάρχουν εσωτερικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν στο κράτος, όποιο και να είναι, να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις διεθνών οργάνων. Αυτό δεν υπάρχει σε πολλά, στα περισσότερα ε, κράτη διεθνώς. Ε, μιλάμε για το Περού, για την Κολομβία, για την Κώστα Ρίκα. Ε, καμία δεν αποτελεί καλό παράδειγμα. Ε, δυστυχώς τα ανώτατα δικαστήρια λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις. Το ανώτατο δικαστήριο του Μεξικού έδρασε εξαιρετικά. Στην ε, περίπτωση της Αργεντινής ε, ελέγχθη από το κράτος ότι δεν δέχεται απόλυτα την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου, αλλά θα την, θα την εφαρμόσει παρόλα αυτά. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν εσωτερικοί μηχανισμοί για την συμμόρφωση, τότε δεν θα υπάρχει συμμόρφωση 100%. Πρόκειται λοιπόν για έναν αμφίδρομο διάλογο, ο οποίος θεσμοθετείται. Θα πρέπει να μιλήσουμε για εσωτερικούς μηχανισμούς που επιβάλλουν τη συμμόρφωση. Και αυτό αφορά και την Ευρώπη και το διαμερικανικό σύστημα και νομίζω ότι με αυτή την παρατήρηση δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Τέλος, χρειαζόμαστε συνεργασία και συντονισμό, γιατί μιλάμε για καθολικές αξίες, μιλάμε για την προάσπιση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη στιγμή που όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά ε, μπορούν να είναι απαιτητά ακόμα και από το τελευταίο φυσικό πρόσωπο επί της γης. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι επιτυγχάνουν και χώρες της Ευρώπης όπως η Ισπανία η Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, και, ε, αναφέρθηκα και στη Νορβηγία που δεν ε, ανήκει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει όλες αυτές οι χώρες έχουν συνεισφέρει και με δικές τους αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους προσκεκλημένους μας για τη συνεισφορά τους και θα μας δώσουμε νομίζω χρήσιμε ιδέες στο Κοινοβούλιο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Στο δε μεσημεριανό έμαθα πως υπάρχουν δύο χώρες τις οποίες δεν αναφέραμε δεν έχουν κυρώσει την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι η ΙΠΑ και ο Καναδάς και ενώ ασχολούμαστε με τις χώρες Λατινικής και της Κεντρικής Αμερικής δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό στις ε, διμερείς μας σχέσεις να τους ε, ζητήσουμε γιατί επί Προέδρου Κάρτερ είχαν σκεφτεί να υπογράψουν και να κερώσουν ε, την συνθήκη και να συνεννοηθούν και με την καναδική κυβέρνηση. Να δούμε τι τους εμποδίζει και αυτούς να υπογράψουν. Ε, δεν ε, μπορώ να σας διώξω, αλλά δυστυχώς πρέπει. Βλέπω πως ο κύριος Ταβάρες έχει νομίζω μια απάντηση για την ε, ερώτηση που είχε κάνει στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. αν πείτε όχι... Α, όχι, είστε έτοιμοι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε σας χαιρετώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους επόμενους εμπειρογνώμονες να έρθουν και εντωμεταξύ έχετε εσείς τον λόγο για να απαντήσετε το ερώτημα για την παράνομη μετανάστευση στο Ισραήλ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάνει λίγο θόρυβο μέσα στην αίθουσα. Τώρα θα γίνω λίγο πιο αυστηρή και παρακαλώ όλοι όσοι δεν ενδιαφέρονται για την απάντηση που θα δοθεί ή να φύγετε από την αίθουσα ή οι υπόλοιποι να καθίσετε. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουν στην Επιτροπή των Σχέσεων με το Ισραήλ προηγουμένως και γι' αυτό δεν μπορούσα να είμαι εδώ παρόν για να απαντήσω. Το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μόλις είδαμε την έγκριση αυτού του νόμου και όταν ακόμη διεξάγονταν ακόμη συζητήσεις ήρθαμε σε επαφή με τους ομολόγους μας στο Ισραήλ διότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας και που είναι και το κέριο σημείο της απάντησης είναι να διαχωρίσουμε αφενός με τις διεθνείς υποχρεώσεις Σύμβαση της Γενέβης, ε, πρωτόκολλα κλπ. Να το διαχωρίσουμε από την απάντηση που μας έδωσαν άμεσα οι Ισραηλινοί που είναι η κυριαρχία ενός κράτους που μπορεί να έχει νομοθεσία για την πρόληψη απειλών ασφαλείας, κυρίως ασφαλείας. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα που θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Και οπωσδήποτε θα το έχουμε στην ημερήσια διάταξη της Υποεπιτροπής ε, που έχουμε με το Ισραήλ που προβλέπεται για το Μάιο για τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάπου τον Απρίλιο-Μάιο το προγραμματίζουμε. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί τόσο άμεσα στην ερώτηση του κυρίου Βουλευτού. Διότι εδώ υπάρχει ένας νόμος του Ισραήλ που εξάλλου υπήρχε ήδη από το 1954 είχε τροποποιηθεί. Ήταν ένας νόμος ε, για την ασφάλεια σε σχέση με την είσοδο στο Ισραηλινό έδαφος και αυτός ο νόμος συνυπήρξε με νόμους για τη μεταχείριση των μεταναστών και των ετούντων άσυλο ε, νόμους που εφαρμόζει το Ισραήλ σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενέβης που έχει επικυρώσει το Ισραήλ. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος ε, εν ονόματι αυτού του νόμου για ε, την ε, ασφάλεια που είναι πιο δεσμευτικός από το προηγούμενο νόμο υπάρχει ο κίνδυνος να παραβιάζονται τα δικαιώματα βάσει της Σύμβασης της Γενέβης. Ευτυχώς το Ισραήλ έχει κυρώσει τη σύμβαση της Γενέβης του 1951 και όλες τις σχετικές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα παρακολουθούμε λοιπόν πολύ προσεκτικά το τι θα γίνει με αυτή την νομοθεσία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται περί παραβίασης της Σύμβασης της Γενέβης όσον αφορά τον νόμο για την ασφάλεια, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μήπως υπάρξει κάποιο ε, γλίστριμα ή κάποιες ε, επικίνδυνες συνέπειες. Ω απάντηση λοιπόν προ τον κύριο Βουλευτή, θέλω να πω ότι το ερώτημα το γνωρίζουμε, το παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά και η απάντηση προ το παρόν είναι ότι οι συμβάσει τι οποίε έχει κυρώσει το Ισραήλ θα τηρηθούν. Σα ευχαριστούμε. Κύριε Ταβάρε. Ευχαριστώ πολύ. Από τις τέσσερις ερωτήσεις που απευθύναμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, απαντήθηκαν οι τρεις. Τι κάνατε και τι θα κάνετε μέχρι το Μάιο, όπως μας είπατε, με αυτή τη συνάντηση που θα έχετε με τις Ισραηλινές αρχές. Και για το πρώτο ερώτημα, ότι ένας νόμος περί ασφαλείας ε, του Ισραήλ δεν είναι αυτός καθεαυτός το πρόβλημα, αλλά η εφαρμογή του νόμου θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της Σύμβασης της Γενέβης. Ένα ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Πώς θα έχουμε κάποια στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή. Ξέρω ότι εγκρίθηκε στις 9 Ιανουαρίου από την ΚΝΕΣΕΤ. αλλά δεν ξέρω σε τι σημείο εφαρμογής αυτού του νόμου βρισκόμαστε. Και θα ήθελα να γνωρίζω αν μπορούμε να έχουμε κάποια παρακολούθηση των γεγονότων επιτόπου από την αντιπροσωπεία μας στο Ισραήλ και αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια γραπτή έκθεση πριν από τη συνεδρίαση του Μαΐου για να μπορούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Επιτροπή. Ναι, βέβαια, Ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Και το σημαντικό δεν είναι ο νόμος, αλλά ο εφαρμοστικός κανονισμός του νόμου και η εφαρμογή του νόμου στην πράξη. Η Σύμβαση της Γενέβης ε, ε, προέχει ε, και εδώ θα πρέπει ε, να δούμε τα θέματα ασφάλεια σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου και τη Σύμβαση τη Γενέβη. Ακριβώ αυτό το οποίο λέτε λοιπόν θα προσπαθήσουμε και εμεί να συνεχίσουμε ε, να εφαρμόζουμε. θέλουμε να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιο μπαίνει στην κατηγορία τρομοκράτη, παραδείγματο χάρη. Αλλά αυτό είναι κάτι που έχει σχέση με τη διαφάνεια που επικρατεί σε κάθε κράτος. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να μην παραβιάζεται η Σύμβαση της Γενέβης του 51 και το δικαίωμα στη μην επαναπροώθηση. Δεν μπορώ να πω τώρα σε λεπτομέρειες λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά ακριβώς το πρόβλημα που έχει το Ισραήλ του ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δέχεται να μπουν στο Ισραήλ και παρισφρίοντας στο Ισραήλ να πλήττεται η ασφάλεια, ε, ακριβώς ε, δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να προστατεύονται τα άτομα τα οποία η Σύμβαση της Γενέβης υπάρχει για να προστατεύει. Και γι' αυτό βρισκόμαστε συνεχώ σε επαφή με το Ισραήλ και θα σα ενημερώσουμε για τη συνέχεια που θα δοθεί. Ο κ. Σταβάρη, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κανονισμό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Όχι. Και σα έχουν δώσει κάποια προθεσμία. Όχι ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρο. Επομένως αυτό το θέμα θα το έχουμε κατ' επανάληψη μέχρι να έχουμε κάποια εξέλιξη. Περνάω τώρα στο σημείο 10, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία. Ένα θέμα ε, στο οποίο θα συμμετέχει και η ε, αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Μαγκρέμπ. Καλώς ήρθατε κύριε Παντσέρη, που είστε πρόεδρος αυτής της επιτροπής, αυτής της αντιπροσωπείας. Και η πολιτική μας στην ε, Ντρουά είναι ότι κάθε σε κάθε συνεδρία θα σας καλούμε. Θα είστε συχνά μαζί μας, κύριε Πανσιάρη, πράγμα που είναι θετικό. Καταλαβαίνω ότι είναι και φόρτος εργασίας για σας, γιατί έχετε πάρα πολλές χώρες στην αντιπροσωπεία σας. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, ιδιαίτερος που ήρθατε. Όπως είπαμε, Κάθε φορά εξετάζουμε μια διαφορετική χώρα. Συγκρίνοντας τις εξελίξεις με το τι έχει γίνει σε άλλες χώρες, η Αλγερία δεν ήταν στο επίκεντρο μέχρι τώρα. Υπήρχαν βέβαια ταραχές στο Αλγέρι, στην πρωτεύουσα, στις αρχές του 2011, αλλά στη συνέχεια, από όσο γνωρίζω, δεν είχαμε μαζικές διαμαρτυρίες στην Αλγερία μέχρι τώρα. Παρ' αυτά, Υπάρχουν διάφορα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία και αυτό θα μας απασχολήσει σήμερα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η Αλγερία έχει κυρώσει διεθνή μέσα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και καλέσαμε πολλούς ε, και έχουμε καλέσει πολλούς ε, παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών για να παρακολουθήσουν την κατάσταση και το Φεβρουάριο του 2011 ήρθε η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ε, που υπήρχε από το 1992 και αυτό είναι θετικό αλλά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στην υποεπιτροπή μας, ε, θέλουμε να εξετάζουμε τα προβλήματα τα οποία παραμένουν ως προς τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε καλέσει λοιπόν εμπειρογνώμονες, τον κύριο Ραμούν, που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αλγερινής Ένωσης ε, Υπεράσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχουμε και τον κύριο Παντσέρη, πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Μαγκρέμπ και τον ε, επικεφαλής της, ε, του τμήματος Μαγκρέμπ στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Φάντη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ και δίνω το λόγο στον κύριο Ραμούν να μας ενημερώσει για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω ότι εκπροσωπώ τρεις οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχουμε μαζί μας ε, τους εκπροσώπους των οικογενειών ε, αγνοωμένων στην Αλγερία και το Συνδικάτο Προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης. Μαζί με τους φίλους μας ε, του Ευρωμεσογειακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίσης συνεργαζόμαστε. Και θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας, αλλά παράλληλα νιώθω και μια πικρία, διότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία. Διότι η κατάσταση, όπως αναφέρατε κι εσείς, δεν είναι λαμπρή, δεν είναι πολύ πιστική η κατάσταση. Και εδώ θέλω να αναφέρω καταρχήν κάποια στοιχεία ανάλυσης και να αναφέρω και το αίτημα που θα διατυπώσουν οι διάφορες οργανώσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω, που αναφέρετε κι εσείς, ε, ε, είναι η άρση ε, της κατάστασης ε, εκτάκτου ανάγκης από τις 23 Φεβρουαρίου του 2011. Αυτή η κατάσταση, αυτή απόφαση ε, δεν προέκυψε από επιθυμία ανοιχτού πνεύματος εκ μέρους ε, του αλγερινού καθεστώτος κατόπιν διαδηλώσεων και κατόπιν αγώνα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προέκυψε. Θεωρούμε ότι είναι ε, τύπης άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, διότι η πρακτική που ακολουθεί το πριν από τις 23 Φεβρουαρίου του 2011 συνεχίζεται και συνεχίζει να υπάρχει βία και καταστολή μετά την άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε αυτή την απόφαση. Τώρα που κοντεύουμε 23 Φεβρουαρίου του 2012, τι απολογισμό μπορούμε να κάνουμε ένα χρόνο μετά την απόφαση άρσης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Σήμερα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δικαίωμα του συνέρχεστε, τι γίνεται με το δικαίωμα της δήλωσης και της διαμαρτυρίας μαζί με συναδέλφους συνεχίζει να υπάρχει περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων. Η οργάνωση SOS Αγνοουμένων κάθε Τετάρτη κάνει μια συνέλευση ζητώντας μεγαλύτερη δικαιοσύνη για τα θέματα των αγνοουμένων. Βλέπουμε ηλικιωμένες γυναίκες και ηλικιωμένους ε, άνδρες μητέρες και πατέρες και αδέρφια των αγνοουμένων. Και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του ότι συνεχίζει να υπάρχει, να ισχύει η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν έχουν το δικαίωμα έκφρασης όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και ακόμη χειρότερα, ε, ακούμε κάποιους εταίρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ε, ακούμε και από το καθεστώς, ότι η Αλγερία δείχνει ανοιχτό πνεύμα, δείχνει κάποια προδιάθεση για άνοιγμα. Και μπορώ να σας το αποδείξω. Το Αλγερινό Κοινοβούλιο ενέκρινε και δημοσίευσε στην επίσημη εφημερίδα τρεις νόμους. Ως διαδικασία και ως σεβασμός προς το Σύνταγμα, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Αλγερίας, ο πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου, που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συνταγματικότητας των ε, νόμων, είχε τη δυνατότητα να εξετάσει αυτού του νόμου εδώ και 7 μήνες και οι δύο δικαστές που ορίστηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από το ίδιο συνταγματικό συμβούλιο εδώ και ένα χρόνο δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για τον νόμο για τη δυνατότητα του συνέχεστε θα σας διαβάσω χάρη παραδείγματος το άρθρο 39 του νόμου σχετικά με την σύσταση ενώσεων. Αναφέρεται η αναστολή δραστηριοτήτων ενώσεων ή διάλυση ενώσεων σε περίπτωση που υπησέρχεται στα εσωτερικά της χώρας. Πραγματικά εν είδη Κάφκα θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει ε, τέτοιου είδους άρθρα. Απαγορεύεται η λειτουργία ενώσεων ε, με αυτό το άρθρο 39, διότι αυτές οι ενώσεις ασχολούνται με τα εσωτερικά της χώρας τους. Τι άλλο θα έκαναν. Επίσης, η, δημιουργία, η διαδικασία δημιουργίας ενώσεων με τον παλαιό νόμο οι ενώσεις θα υπόκειταν σε κάποιο καθεστώς δηλώσεων. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνουν τη δήλωση τα μέλη και θα ε, λάμβαναν ε, απόδειξη υποβολής της αιτήσεως και θα μπορούσε να εγκριθεί η σύσταση οργάνωσης. Ενώ ε, τώρα δεν έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα. Αυτά σας τα αναφέρω ως παράδειγμα γιατί βασίζονται σε κάποια άρθρα του νέου νόμου για τις ε, οργανώσεις και ενώσεις. Ο νόμος για τα πολιτικά κόμματα ε, και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το γενικό κλίμα που ισχύει στη χώρα μετά την περίφημη άρση της απόφασης, άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Υπάρχει απόφαση η οποία δίνει περισσότερες εξουσίες στον Υπουργό Εσωτερικών και θέτει όρους στα πολιτικά κόμματα και στις δραστηριότητές τους. Δηλαδή, δεν υφίσταται η δημοκρατία ως τρόπος λειτουργίας και ως τρόπος άσκησης των ε, διαδικασιών του κράτους επιβάλλονται στα κόμματα αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουν. τρίτος νόμος, ο νόμος για την ε, πληροφόρηση. Το άρθρο 2 του νόμου αυτού θα σας το διαβάσω. Η πληροφόρηση είναι μια δραστηριότητα που ασκείται ελεύθερα στο πλαίσιο του παρόντος οργανικού νόμου. Θα πρέπει να τηρείται το Σύνταγμα και οι νόμοι της Δημοκρατίας το μουσουλμανικό θρήσκευμα και οι άλλες θρησκείες, η εθνική ταυτότητα και ε, οι πολιτιστικές αξίες της, της ε, κοινωνίας, οι απαιτήσει ασφαλείας και εθνικής άμυνας, οι απαιτήσει δημόσιας τάξης, τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, οι υποχρεώσεις ε, του δημοσίου τομέα και ο, πληροφορεί, ο πολίτης θα πρέπει να πληροφορείται λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα θέματα όπως επίσης και την τήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της συλλογική αξιοπρέπειας. Δηλαδή, η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία των δημοσιογράφων υπόκειται σε όλα αυτά. Θα πρέπει μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις να ασκείται η ελευθερία του τύπου. Τα μέσα ενημέρωσης λοιπόν είναι ελεγχόμενα, είναι υπό αυστηρό έλεγχο από το τμήμα ασφάλειας, το DRS. Όταν αναφέρεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης μιας χώρας και η νομιμότητα μιας χώρας εσωτερικά και εξωτερικά, από τις ε, επισκέψεις σας και από την αντιπροσωπεία σας στην Αλγερία θεωρείτε ότι υπάρχει ε, νομιμότητα της κυβέρνησης. Τα ε, εθνικά θέματα αποφασίζονται έξω από τα θεσμικά όργανα του κράτους. Αυτό το όργανο, το DRS, έχει εξαιρετικές εξουσίες, εξουσίες ε, που συνδέονται και με την τρομοκρατία και με τη διαχείριση ε, του θέματος των αγνοουμένων ε, και ασκείται εκβιασμός στις οικογένειες των αγνοουμένων να υπογράψουν το έντυπο που δηλώνει τον θάνατο των οικείων τους έναντι χρημάτων. Είναι τρέχουσα πρακτική στην Αλγερία αυτός ο εκβιασμός. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλγερίας, λυπούμεθα την ε, απουσία σαφούς θέσεως για την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία. Και αυτό είναι κάτι που προκύπτει από τις δευτεριότητες των οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών επιτόπου. Μετά την ε, Αραβική Άνοιξη, η πολιτική γειτονίας θα πρέπει να δώσει καρπούς, να δείξει ότι επιτέλους καταλάβαμε και πρέπει να αλλάξει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Μεσογείου και των χωρών του Μαγκρέμπ. Κάνουμε έκκληση λοιπόν σήμερα. Αυτή η νέα πολιτική να ερμηνευθεί στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλγερίας και να μην περιορίζεται μόνο σε οικονομικά θέματα στις σχέσεις αυτές. Η αναγνώριση της κοινωνίας των πολιτών στην Αλγερία, που θα πρέπει να είναι αυτόνομη, είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται για όλους μας. Και σε αυτό το πλαίσιο και με αυτή την προοπτική, η βούληση ε, της Αλγερίας να συνεργαστεί και ε, να ε, οργανώσει τις, νομοθετικές, τις βουλευτικές εκλογές πιστεύω ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία διότι όλα αυτά τα στοιχεία που απαριθμίσαμε μας οδηγούν στο να πούμε ότι σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές έχουμε ένα ραντεβού με την ιστορία. Πώς θα διεξαχθούν αυτές οι εκλογές. Οι εγγυήσει που διατυπώνονται από το Αλγέρι σχετικά με την ε, σωστή διεξαγωγή των εκλογών θα τηρηθούν ζητούμε μια σαφή δήλωση σχετικά με την υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία και ζητούμε μια ανοιχτή συζήτηση παρουσία της ε, Λεβισάστον, το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς και ακριβείς θέσεις που θα εκφραστούν εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, συγκεκριμένες προτάσεις σας και για το ότι υπογραμμίσατε ξανά το πόσο σοβαρές ήταν οι περιπτώσεις των εξαφανίσεων από, την, από τον καιρό του πολέμου νομίζω ήδη του εμφυλίου και η κατάσταση τότε ήταν πολύ στα ΜΜΕ αλλά μετά όταν περνάει λίγο χρόνο ξέρετε, ξεχνιούνται αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας τα υπενθυμίσατε και για το ότι βοηθάτε και μας λέτε πως ε, οι συγγενείς ε, των θυμάτων, των εξαφανισμένων ε, εξακολουθούν να θέλουν να μάθουν τι απέγιναν οι οικοί τους. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Φάντι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μας πείτε τι κάνετε εσείς ως προς αυτό όχι τόσο πολύ να μας πείτε το τι έχει κυρώσει η Αλγερία. Ε, υποθέτω δηλαδή πως η Αλγερία δεν έχει υπογράψει την συνθήκη περί... τη σύμβαση περί εξαφανίσεων. Αλλά πείτε μας ε, κατά πόσο συζητάτε το ζήτημα αυτό. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ και και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να απαντήσω επί του θέματος. Θα ήθελα να πω ότι ακούσαμε με μεγάλη προσοχή αυτά που μας είπε ο εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών και παρακολουθούμε εκ της σύνεγγης την κατάσταση στη χώρα για να, έχουμε, για να προωθήσουμε έναν διάλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής. Πρώτον, η πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για να αποστείλει ε, παρατηρητές για τις εκλογές, διενέργεια εκλογών του Μαΐου του 2012. Μία διερευνητική αποστολή θα μεταβεί από τις 31 Ιανουαρίου για να δούμε πώς μπορεί να ε, αποσταλεί αυτή η ομάδα παρατηρητών. Πρόκειται για μία επίσκεψη ρουτίνας, δηλαδή καταρχήν υπάρχει ε, αποστέλλεται μία διερευνητική επιτροπή, υπάρχει η θέληση. Η κυρία ε, Άστον απάντησε στον Υπουργό Εξωτερικών και εάν πληρούνται οι όροι θα ε, αποστείλουμε παρατηρητές. Ένα άλλο θέμα είναι το ότι από το 11 και μετά ε, έχουμε έναν διάλογο με την Αλγερία ή για θέματα ασφάλειας και ε, προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό γίνεται από το 2011 και μετά και αυτό γίνεται και μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης για να ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, θέματα διακυβέρνησης και κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να προωθήσουμε το διάλογο αυτό με την Αλγερία πέρα από τις άτυπες επαφές μας. Και το τρίτο στοιχείο είναι η πρόσφατη απόφαση της Αλγερίας να δεχτεί την ευρωπαϊκή πολιτική γυτνίασης και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αρχίζει το διάλογο επί του θέματος για να προβλέψει ένα πρόγραμμα δράσης στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Ένα σχέδιο δράσης θα μας επιτρέψει να ορίσουμε καλύτερα τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κατάστασης ε, ε, και της κατάστασης δικαίου. Μια πρώτη άτυπη συνάντηση θα γίνει με τις αλγερινές αρχές και θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο έτσι ώστε να ορίσουμε αυτό το σχέδιο δράσης. Σχέδιο δράσης μετά την αλλαγή της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2011 και στόχος μας είναι να διαβλέψουμε συγκεκριμένους στόχους με δίκτες αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε να έχουμε έναν διάλογο με βάση απτά στοιχεία. Θεωρούμε ότι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι ύψης της σημασίας και θα θέλαμε η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει σε αυτό το σχέδιο δράσης. Και αυτό το διαβιβάσαμε στην ε, κυβέρνηση της Αλγερίας. Αυτά είναι τα στοιχεία προς το παρόν. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα. Thank you, Mr. Fanti. Ευχαριστούμε κύριε Φάντη. Ο κύριος Παντσέρη έχει το λόγο τώρα από την αντιπροσωπεία του Μαγκρέβ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αλγερία έχει ορισμένα ζητήματα προς αντιμετώπιση γιατί ζει σε μία αντίφαση. Είναι γεγονός ότι έχει έναν πολύ καλό έλεγχο ως προς την υπεράσπαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρόλα αυτά δεν υπάρχει συνοχή στη νομοθετική διαδικασία έτσι ώστε να συμβαδίζει με αυτή τη στη γραμμή, με αυτή την επικυρωτική διαδικασία δηλαδή. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να πούμε στεναρά ότι είναι μια χώρα που θα πρέπει να εφαρμόσει ένα πιο προωθημένο πρόγραμμα εκδημοκρατισμού μέσα στα πλαίσια του πολιτικού πλουραλισμού, του ενωσιακού ε, πλουραλισμού και τη συμμετοχής των συλλογικών φορέων. Αυτό θα πρέπει να δούμε και στις σχέσεις μας, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλγερίας, μέσα στα πλαίσια της νέας πολιτικής γειτονίας. Γιατί με αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο υπό οικονομικούς όρους. Υπάρχουν ε, δις δολαρίων που προέρχονται από τον τομέα της ενέργειας. Γίνονται πωλήσει σε πολλές χώρες, γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε σε επίπεδο σύνδεσης και εδώ να είμαστε πιο διεκδικητικοί, έτσι ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να ε, συνδεθούν με αυτό το πλαίσιο πιο αποφασιστικά. Αυτό το είπαμε και πρόσφατα πρόσφατα στο Αλγέρι στις συναντήσεις μας, όπου προβάλαμε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή να προωθήσουμε μια ε, μεγάλη συνεργασία, αλλά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών είναι ύψης της σημασίας ε, για εμάς. Ως προς το θέμα του παρατηρητηρίου της διενέργειας εκλογών, θα ήθελα να πω στον κύριο Ραμούμπ αυτά που ε, αφορούν και όσα προανέφερε ο κύριος ε, Φάντη. Εμείς ζητήσαμε την αποστολή ομάδας παρατηρητών. Αυτό το ζητήσαμε όταν μεταβήκαμε στην Αλγερία για να αποφύγουμε κάτι το οποίο ήταν λανθασμένο στο παρελθόν. Όταν διενεργούνται εκλογές συμμετείχαν διάφοροι ευρωβουλευτές, φίλοι της Αλγερίας, φίλοι του Τάδε του Δίνα, επισφραγίζοντας την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις ε, εκλογικές διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η σφραγίδα να είναι και επίσημη. Το λέω για ότι ίσως να μην υπάρξει αποστολή παρατηρητών διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάντε εσείς την αξιολόγηση, λέω προς την Κομισιόν, το πρότυπό μας το εκπονήσαμε στην Τινησία, στην ομάδα παρατηρητών που απεστάλλει. Μιλάμε για πλήρη διαφάνεια, ίσες ε, διαδικασίες ε, δικαιοσύνης στους όρους πρόσβασης και θεωρούμε ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού πλήρως εάν ε, δεν πληρούνται με βάση τις συναντήσεις που θα γίνουν στο εγγύς μέλλον ας το πούμε ε, δημοσία ότι δεν θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να ε, είμαστε αδιάλακτοι έτσι ώστε να είμαστε αξιόπιστοι και να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε εκεί για να πούμε τη δική μας ε, άποψη, γιατί τασόμαστε υπέρ της διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Παντσέρη για τις δηλώσεις σας για τις εκλογές αλλά και για το ότι είπατε πως στη μελλοντική συμφωνία με την Αλγερία τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο από το παρελθόν. Ενθαρρυντικό αυτό. Λοιπόν, στον καταλογό μου τώρα είναι η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ραμόν για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Και να πω ότι η κατάσταση της Αλγερίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ε, μία κατάσταση δυσχεριών για μας. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Αλγερία γιατί καταρχήν τη στιγμή που θα προκηρυχθούν εκλογές με νόμους που δεν συνάδουν με τις με δημοκρατικές διαδικασίες για μας αυτή είναι μια προτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών που βασίζεται σε κατασταλτικά άρθρα του συντάγματος. Δεν είναι όπως την Τίνιδα, όπου ένας ανεξάρτητος, ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών έπρεπε να διοργανώσει τις εκλογές. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για να δούμε κατά πόσο ε, υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει μία εναλλαγή, δηλαδή εάν αλλάξει σκητάλη στην εξουσία. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα Ισλαμικό κόμμα το οποίο ε, φιλοδοξεί να μαζέψει τις ψήφους που ίσως θα χάσει η τωρινή κυβέρνηση. Ποια όμως είναι η πραγματική κατάσταση του λαού. Το θέμα για μας τους ευρωβουλευτές είναι ότι δεν έχουμε συνομιλητές ούτε στο κοινοβούλιο σας, ούτε στην ε, κοινωνία σας, στην πολιτική κοινωνία. Δεν έχουμε συνομιλητές γιατί δεν είναι το ίδιο να ανήκει κανείς στην κοινωνία των πολιτών και ενός πολιτικού κόμματος που εκπροσωπεί την αντιπολίτευση εκεί. Εμείς δεν γνωρίζουμε ένα πολιτικό κόμμα με δημοκρατικές φιλοδοξίες που να βρίσκεται εδώ έτσι ώστε να είναι συνομιλητής μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να προωθήσουμε διάλογο. Ούτε μπορούμε να κάνουμε, ούτε μπορούμε να υποκαταστήσουμε την αντιπολίτευση της Αλγερίας. Μπορούμε να βοηθήσουμε την αντιπολίτευση της Αλγερίας, αλλά δεν μπορούμε να την υποκαταστήσουμε. Και αυτή η αντιπολίτευση πρέπει να είναι καλώς διαρθρωμένη, να είναι οργανωμένη. Δεν χρειαζόμαστε καταγγελίες άρθρων. Θα πρέπει να υπάρχει μία λαϊκή κινητοποίηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε στο αίτημά σας αυτό. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει εδώ το αίτημα αυτό. Και επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα που αναχαιτίζουν την άσκηση ε, δικαιωμάτων και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα θέλαμε να εξαφανιστούν αυτά τα άρθρα ή νόμοι, έτσι ώστε να ανακύψει μία πραγματική δημοκρατία και αυτή η καταγγελία μπορεί να τύχει της υποστήριξής μας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την οικοδόμηση της δημοκρατίας. Μπορούμε να καταγγείλουμε και να πούμε ότι δεν πληρούνται οι όροι για να υπάρξει μία εναλλαγή στην εξουσία. Και η Κομισιόν έχει προβεί στη σύσταση μίας υποεπιτροπής, αλλά δεν ξέρουμε με ποιον. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα θέματα συζήτησης. γιατί θα πρέπει να δούμε κατά πόσο συμμεριζόμαστε ή όχι τις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Αλγερίας. Θα πρέπει να ε, διαγραφούν αυτά τα άρθρα και να ισχύουν οι δημοκρατικές αρχές. Διαφορετικά δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Ρωμέρο. Τώρα θα μιλήσω και εγώ. Έχω ένα ερώτημα. Κύριε Φάντη. Ο κύριος Ραμόν περιέγραψε σε πολλές περιπτώσεις το εξής. Οι προσθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε πρόκειται για ένα σύλλογο είτε είναι συγγενείς που ζητάνε να μάθουν τι έγινε οι οικοί Νομίζω πως όλα αυτά είναι ζητήματα ευρασιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πολιτική λοιπόν της υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι πως σε κάθε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει κάποιος για να στηρίζει το έργο των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πρώτα απ' όλα εάν στην αντιπροσωπεία στο Αλγέρι υπάρχει κάποιος και πόσο εντατικά ασχολείται με την στήριξη των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί καταλαβαίνω από την πρόσφατη ιστορία και την καταπίεση που υπάρχει εκεί πως είναι δύσκολη η δουλειά αυτή γιατί διακινδυνεύονται πάρα πολλά η σωματική ακαιρεότητα οι ανθρωποί δέρνονται και η μνήμη της βίας ε, πριν από λίγα χρόνια με τις εξαφανίσεις θα υπάρχει οπωσδήποτε στην κοινωνία. Δεν είναι κάτι το εύκολο. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένα να μας πείτε το πώς εντατικά εργάζεστε για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Άλλες ερωτήσεις, όχι. Μετά κατόπιν ε, τον κύριο Φάντη θα ήθελα να δώσω λόγο σε εσά ξανά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά με την ερώτησή σας, δεν έχουμε ακόμη μια τοπική στρατηγική στην Αλγερία όσον αφορά τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να προκύψει από μια εργασία όλων των κρατών μελών που βρίσκονται επί τόπου με συνένεση και θα επιδιώξουμε τη δημιουργία μιας στρατηγικής επιτόπου και να ορίσουμε και ένα σημείο επαφής. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες, αλλά όπως κάνουμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία μιας τοπικής στρατηγικής είναι μία από τις στρατηγικές, ένα από τα βήματα που πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο της πολιτικής προσέγγισης με την Αλγερία στις συζητήσεις μας για τα θέματα αυτά. Και θα ήθελα να προσθέσω και μια διευκρίνηση σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Ρομέρο για την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Πολιτικό Διάλογο. Σε όλες τις περιπτώσεις, για όλες τις χώρες εταίρους, αυτές οι υποεπιτροπές δημιουργούνται στο πλαίσιο συμφωνιών σύνδεσης, δημιουργούνται από το Συμβούλιο Σύνδεσης και ο συνομιλητής είναι η κυβέρνηση. Αυτές οι υποεπιτροπές υπάρχουν ακριβώς για να δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει διάλογο με τις κυβερνήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διακυβέρνηση και επομένως ε, να φύγει αυτά τα συγκεκριμένα θέματα κατά τη συζήτηση. Βέβαια, παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αντιπροσωπιών ή μέσω άλλων μέσων μπορεί να έχει διαβουλεύσεις ή επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Αλλά περισσότερο με άτυπο χαρακτήρα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ακόμη. Αυτή, αυτός ο πρώτος διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλγερίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ε, θα δώσει κάποια συμπεράσματα τα οποία θα συζητηθούν εδώ ε, στην Επιτροπή μας. Αλλά θα ήθελα να μου διευκρινίσετε ότι δεν υπάρχει στην Αλγερία, στην αντιπροσωπεία κάποιος που να είναι υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι στρατηγικές η στρατηγική χώρα για την Αλγερία είναι κάτι που το επεξεργάζεστε. Αλλά δεν υπάρχει ένα άτομο που να είναι το άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή ακριβώς για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι παλαιό το αίτημα αυτό. Ο κύριος Φάντη, υπάρχει κάποιος που ασχολείται με το θέμα των ε, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ο πολιτικός μας σύμβουλος ε, στο Αλγέρι. Αυτό που εννοούσα είναι ότι δεν έχουμε ακόμη τοπική στρατηγική, αλλά και βέβαια υπάρχει ένα άτομο που δουλεύει πάνω σε αυτά τα θέματα. Ε, θετικό αυτό και ελπίζω ότι και η κοινωνία των πολιτών ε, και όλοι οι προασπίζοντες στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία θα υποστηρίζονται από την αντιπροσωπεία οποτεδήποτε το χρειάζονται. Κύριε Ραμούν, θέλετε να συνοψίσετε. Σας ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι για τις παρεμβάσεις που ακούσαμε από τον κύριο Παντσέρη, τον κύριο Φάντη και την κύριο Ρομέρο διότι μου επιβεβαιώνουν, ε, υπάρχουν διαπιστώσεις που και οι τρεις ομιλητές ε, επιβεβαιώνουν. Είναι σαφές ότι η Αλγερία είναι μια χώρα που έχει υπογράψει σχεδόν όλες τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις, όπως είπε ο κ. Παντσέρη. Όμως ισχύει επίσης ότι αυτά τα νομικά κείμενα ε, αυτά τα νομοθετικά κείμενα που σας ανέφερα δεν είναι συμβατά με τα διεθνή κείμενα που έχει κυρώσει η Αλγερία και χαίρομαι που το ακούω και από εσά. Δεύτερον, όσον αφορά την αντιπροσωπεία στο Αλγέρι, κάθε φορά μας κάνει εντύπωση το πώς χειρίζεται τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η SOS Αγνοούμενη, που είναι πολύ δραστήρια οργάνωση επιτόπου, ποτέ δεν παίρνει πρόσκληση από την αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποτέ δεν έχει ακούσει την άποψη αυτής της οργάνωσης και είναι κρίμα. Στην Αλγερία έχουμε ένα σύστημα που ονομάζεται σύστημα κλώνων, όπως το αποκαλούν οι συνδικαλιστές. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα αυτόνομο συνδικάτο στη δράση του, το καθεστώς δημιουργεί άλλο ένα συνδικάτο με το ίδιο όνομα. και όταν η αντιπροσωπεία καλεί τα συνδικάτα που έχουν το όνομα ΣΝΑΠΑΠ, είναι πολλά τα συνδικάτα με το ίδιο όνομα, ακριβώς για να μποϊκοτάρει τη δράση του συνδικάτου. Ε, είναι μια αρχή του καθεστώτος. Θυμάμαι κατά τη δεκαετία του 1990 μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού ήταν οι επισκέψεις ε, της αντιπροσωπείας στην Αλγερία ή ευρωβουλευτών στην Αλγερία. Ήμασταν απομονωμένοι, δεν είχαμε υποστήριξη. Από το 1991 η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες της Αλγερίας πάντοτε προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν την ε, διεθνή κοινή γνώμη. Σχεδόν εννέα φορές έχουν γίνει εκλογές από το 1991 και μετά. Το 95 προεδρικές, το 97 βουλευτικές, το 99 προεδρικές, 2002-2007 βουλευτικές, 2004 προεδρικές, 2009 προεδρικές, 2012 βουλευτικές και δημοτικές. Αυτή η διαδικασία επέτρεψε τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Όχι είναι η απάντηση. Είχαμε πέντε προέδρους, πέντε συντάγματα. Αλλά κανένα σύνταγμα δεν προστάτευε τον πρόεδρο. Ένας πρόεδρος δολοφονήθηκε, ένας παρετήθηκε, ένας οθήθηκε στην παρέτηση, ένας δολοφονήθηκε και ο τελευταίος πρόεδρος θέλει να μείνει ισόβια πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της Αλγερίας πέραν από δημοκρατικούς κανόνες, και έξω από την εξουσία των θεσμικών οργάνων στην Αλγερία. Δεν μπορεί να προχωρήσει προς ένα άνοιγμα της χώρας αυτή η κατάσταση. Ε, τώρα αλλάζει η κατάσταση στις χώρες του Μαγκρέμπ και αλλάζει η αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες αυτές. Ε, ακριβώς αυτό το οποίο κάνετε, το ότι τονίζετε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, στις συναντήσεις που κάνετε στο πλαίσιο της πολιτικής ε, γειτονίας είναι ένα σημαντικό βήμα από δική σας πλευράς. Οι χώρες του Μαγκρέμπ έκαναν την επανάστασή τους και τώρα πρέπει να κάνετε και εσείς την επανάστασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Um, σα ευχαριστούμε. Νομίζω πως ε, η παρατήρησή σα πως η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επαφή με κάποιες μόνο ΜΚΟ ε, ακούστηκε και νομίζω πως αυτό ισχύει όχι μόνο στην Αλγερία ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί για το ποιος είναι πραγματική μοικείο. Δεν ελέγχεται αυτό εύκολο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από όσο γνωρίζω, νομίζω πριν από έξι χρόνια, κύριε Παντσέρη, γιατί είμαι καινούργια εγώ, μου το είπαν τώρα μόλις, πριν από έξι-εφτά χρόνια υπήρχε το τελευταίο ψήφισμα που πέρασε για την κατάσταση στην Αλγερία Οπότε πρέπει να σκεφτούμε το γιατί. Και να δούμε αν έχει προσθέμενη αξία ένα νέο ψήφισμα για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εκλογέ είναι άλλο θέμα. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη, να δούμε πώς μπορούμε να σας στηρίξουμε καλύτερα. Ο κύριος Φάντη τώρα ήθελε το λόγο για το θέμα των ΜΚΟ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, για να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα σημειώνω την δυσαρέσκεια που υπάρχει όσον αφορά τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Εγώ δεν συμφωνώ πλήρως, δεν νομίζω πως η αντιπροσωπεία μας αρνείται να δεχτεί ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα την SOS Disparu, πράγματι υπήρξε μια συνάντηση με τον πολιτικό μας σύμβουλο και τον εκπρόσωπο της οργάνωσης αυτής στο Αλγέρι και είχε προσκληθεί ε, σε μια συνάντηση πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής σας, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Έτσι για να ξέρουμε τα γεγονότα. Το σημειώνω, εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσω με τους συναδέλφους μας για θα τους πω πως υπάρχουν υψηλέ προσδοκίες για ενίσχυση των επαφών. Θα ήθελα επίσης να πω, έχοντα ακούσει τον εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, πως εγώ δεν είπα πως η νομοθεσία της Αλγερίας δεν συμμορφώνεται με τις διεθνείς συνθήκες και θα ήθελα αυτό να γραφτεί στα πρακτικά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όμως, από ό,τι βλέπω, κύριε Φάντη, πρέπει να δουλέψετε λίγο καλύτερα με την αντιπροσωπεία. Βρείτε τους τρόπους. Αλλά νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν τέλος είναι γεγονός ότι το τελευταίο ψήφισμα συντάχθηκε αρκετά χρόνια πριν και οι σχέσεις με την Αλγερία είχαν σταματήσει το 2005, αποκαταστάθηκαν πρόσφατα. Και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα ψήφισμα για τη σύνταξή του, όπου να φαίνεται ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την Αλγερία στα πλαίσια των ε, μεταρρυθμίσεων και να βρούμε τη, τις διάφορες φάσεις, τα διάφορα ορόσημα. Αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. For uh, Βεβαίως, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση για την Αλγερία Είμαι σίγουρος κύριε Παντσέρη πως θα μεταφέρετε τα όσα είπαμε σε αυτή την ομάδα για την παρακολούθηση, την εταιρική σχέση με την νότια γειτονιά μας γιατί υπάρχει μία μόνιμη συζήτηση και νομίζω πως εγώ δεν, δεν ήμουν εγώ στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις αλλά νομίζω πως έδωσαν πάρος στην Αλγερία. Όχι, δεν ξέρω, δεν ήμουνα. Εμείς στην Επιτροπή λοιπόν Ντροά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με ένα μελλοντικό ψήφισμα. Οπότε νομίζω πως τελείωσε η συνεδρίασή μας. Υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Όχι. Οπότε να σας ανακοινώσω πως η επόμενη συνεδρίαση είναι σε 9 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.